Καλό απόγευμα σε όλους. Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι βουλευτέ των Εθνικών Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Τιούτου. Μαζευτήκαμε εδώ απόψε σε αυτή την κοινή διακοινοβουλευτική συνάντηση για το θέμα του ρόλου της Ευρωδίκ και Ευρωάστα καθώς και του Frontex. Σας καλωσορίζω. Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεστε σε τέτοια συνάντηση. Ο συνδυασμός των μελών από τις βουλές των, των χωρών με τους βουλευτές του Ευρωκοινοβουλίου με σκοπό να ασχοληθούμε με το θέμα της οικοδόμησης του Ευρωπαϊκού Χώρου Ελευθερίας, Ασφαλείας και Δικαιοσύνης. Όπως λέει η συνθήκη της Λισαβόνας είναι το θέμα μας. Πέρασαν δύο χρόνια από τότε που τέθηκε σε ισχύ και είπαμε ότι ήταν πολύ σημαντικό ότι επιτέλους ξεκαθαρίστηκε ότι οι πολίτες είναι, βρίσκονται στην καρδιά της ευρωπαϊκής διαδικασίας, της ευρωπαϊκής οικοδόμησης, του ευρωπαϊκού οράματος όπως λέμε και άρα στην καρδιά όλων μας των προγραμμάτων και των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Τιούτου. Δεν έχουμε όμως αρκετά τονίσει πώς τον τρόπο με τον οποίο η νέα αυτή θεσμική διευθέτηση θα εφαρμοζόταν. Λέγαμε πιο παλιά ότι η συνθήκη της Λισαβόνας στόχευε στην απλοποίηση. Αυτό δεν ήταν απόλυτα αλήθεια. Φευσικά ήταν και αυτό αλήθεια, αλλά δεν ήταν η μόνη αλήθεια. Γιατί σε ορισμένα θέματα μπορεί η συνθήκη να καταστήσει τη ζωή των κοινοβουλίων πιο δύσκολη και των εθνικών και του ευρωπαϊκού. Για τον απλό λόγο ότι πρέπει παραπάνω από ποτέ να συνεργαζόμαστε για να ενδυναμώσουμε τα προγράμματα, τα ενωσιακά προγράμματα που αφορούν την ελευθερία, τη δικαιοσύνη και την ασφάλεια. Θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πολιτών όπως τα εξωτερικά σύνορα, την ελεύθερη διακίνηση, στον κοινό μας χώρο καταπολέμηση του διαμεθοριακού εγκλήματος δικαστική και αστυνομική συνεργασία για την καταπολέμηση σοβαρών εγκλημάτων απειλές που μας είναι κοινέ, δουλεμπόριο διαφθορά και δωροδοκία ναρκωτικά, ξέπλυμα βρωμίκου χρήματος ασφάλεια όλοι αυτοί είναι κοινοί μας στόχοι πολέμηση της τρομοκρατίας η οικοδόμηση αυτού του χώρου ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών με τα δικαιώματά τους, με τα πλήρη τους δικαιώματα είναι ακριβώς το θέμα που μας απασχολεί. Γι' αυτό πρέπει να συνεργαζόμαστε ως εθνικοί και ευρωπαϊκοί νομοθέτες όπως προβλέπει το άρθρο 12 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το οποίο σας υπενθυμίζω τα εθνικά κοινοβούλια συνεισφέρουν ενεργά στην εύρυθμη λειτουργία της Ένωσης συμμετέχοντας στην οικοδόμηση του χώρου ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφαλείας για την εφαρμογή όλων των σχετικών κοινοτικών προγραμμάτων. Και σύμφωνα με το άρθρο 70 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αξιολόγηση της Ευρωπόλ και της Ευρωάστα είναι επίσης δικαιοδοσία των Εθνικών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα α 88 και 85. Για όλους αυτούς τους λόγους είχε γίνει η πρώτη διακοινοβουλευτική διάσκεψή μας και τώρα αρχίζει η δεύτερη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο συνεργασίας η πρόεδροι των Εθνικών Κοινοβουλίων στη Στοκχόλμη το 2010 το είχαν πρώτο αποφασίσει και οι πρόεδροι αυτοί είχαν ζητήσει από την τότε Βελγική Προεδρία να υποβάλει προτάσεις για να προγραμματίσει τακτικές συναντήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με εκπροσώπους των Εθνικών για θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών. Αυτό κάναμε λοιπόν και εμείς από τότε και γι' αυτό και γι' αυτό θέλουμε να αυξήσουμε την προστασία των πολιτών μέσω αυτής της συνεργασίας βάσει του ενωσιακού δικαίου. Είναι πρόκληση για τους νομοθέτες, για τη διατήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και το σεβασμό του σε ολόκληρη την Ένωση και για τη διατήρηση των εθνικών νομικών τάξεων και δικαστικών τάξεων. Σύμφωνα με το άρθρο 87 της Συνθήκης της Ένωσης που μιλάει για τις αρχές της αναλογικότητας και της επικουρικότητας ε, πλήρης δηλαδή συμμετοχή και των εθνικών νομοθετών. Όλα αυτά θέτουν ορισμένες προκλήσεις και καθήκοντα που πρέπει να εφαρμόσουμε. Υπάρχουν ορισμένες ευρωπαϊκές υπηρεσίες, το Frontex, το SIPOL, το IASO, ENISA, και η Ευρωπόλ και η Ευρωτζάστ. Υπάρχουν και διακανονισμοί όπως το σύστημα πληροφόρησης του Σέγγεν, το Ευρωδάκ και μηχανισμοί καθώς και ό,τι έχει προβλεφθεί για την ανταλλαγή πληροφοριών. Σιγά σιγά αυτά τα κοινά εργαλεία αρχίζουν να λειτουργούν Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφίσαμε επί της τελευταίας απόφασης του Συμβουλίου για την Ευρωάστ και την Ευρωδίκα και ζητήσαμε από την Κομισιόν τον Σεπτέμβριο του 10 να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις που να πλαισιώνουν τουλάχιστον την κοινοβουλευτική εποπτεία σύμφωνα με το άρθρο 70 της συνθήκης είναι καθήκον του και δικαίωμά του να κάνει αυτή την εποπτεία. Βάσει λοιπόν του χρονοδιαγράμματος που σκοπό είχε να λισαβονοποιήσει τον πρώην τρίτο πυλώνα, έχουμε σημειώσει κάποια καθυστέρηση. Πρέπει να κάνουμε πολλά λοιπόν για να τη γεφυρώσουμε, να την αντιμετωπίσουμε. Αν θέλουμε να εφαρμόσουμε τους στόχους μας με βάση τις προσδοκίες και ελπίδες των πολιτών που εκπροσωπούμε και στα εθνικά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χρειαζόταν λοιπόν να οικοδομηθεί ένας χώρο συνεργασίας των Ευρωβουλευτών και των εισηγητών του Κοινοβουλίου μας με τα, με τα εθνικά Αυτή είναι η λογική που εφαρμόζουμε εδώ. Αυτό είναι, αυτός είναι ο δρόμος που θα ακολουθήσουμε μέχρι να εφαρμοστούν οι στόχοι. Και είναι μεγάλη μας τιμή που σας βλέπουμε σήμερα εδώ. 43 εθνικούς βουλευτές από 25 εθνικά κοινοβούλια. από τουλάχιστον 18 χώρες μέλη. Thank you for bothering. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν. Γνωρίζουμε τη σημασία που έχουν όλα αυτά και θα συμμεριστούμε στην Προεδρία της εκδήλωσης αυτής με την Επίτροπο και Μάλστρομ που είναι υπεύθυνη για τα εσωτερικά καθώς και τον κύριο Γκραμπάτσκι που θα, τον Υπουργό Γκραμπάτσκι που εκπροσωπεί την Προεδρία του Συμβουλίου εξ ονόματος της Πολωνικής Προεδρίας. Πρώτα θα μας μιλήσει η Επίτροπος Μάλστρομ, μετά ο κύριος Ραπάτσκι και θα ακούσουμε και ορισμένες ομιλίες που έχουν υποβληθεί για συγκεκριμένα θέματα και φυσικά θα υπάρξει και συζήτηση φυσικά. Αλλά για να σεβαστούμε το χρονοδιάγραμμά μας δύο μέλη από εθνικά κοινοβούλια και μετά ένα μέλος του Ευρωκοινοβουλίου. Και όλοι, όλοι και όλες θα περιορίζονται σε δύο λεπτά. Δύο λεπτά. Λίγο ευέλικτα, αλλά δύο λεπτά βασικά. Γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι είμαστε αρκετοί εδώ και αρκετές και αν θέλουμε να μιλήσουν όλοι και να εφαρμόσουμε και την ημερήσια διάταξή μας χρειάζεται αυτό το όριο. Σας ευχαριστώ. Τώρα η Επίτροπος Μάλστρομ δέ χωρίς όριο εκείνη. Δεν εφαρμόζεται σε εσά το όριο κυρία Μάλστρομ, εσείς μπορείτε να πείτε ό,τι και όσα θέλετε. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι. Είμαι ε, πολύ... Ε, ε, αισθάνομαι ότι με τιμάτε που με καλέσατε σήμερα και είστε τόσο πολλοί για να συζητήσουμε αυτό το θέμα και έχετε ταξιδέψει από πολύ μακριά. Θα συζητήσουμε λοιπόν σήμερα και αύριο, διότι η ασφάλεια είναι προτεραιότητα για τους πολίτες. Όποτε γίνεται ένα ερωτηματολόγιο και αναρωτιόμαστε ποια είναι τα δικαιώματα που είναι βασικά για τους πολίτες η ασφάλεια είναι πάντα πολύ υψηλά. Πρέπει να ζουν σε μία ασφαλή περιοχή και να χαίρουν των δικαιωμάτων τους ότι ε, θα έχουν ιδιωτική ζωή και ότι θα μπορούν να προστατεύουν και τα ιδιωτικά τους δεδομένα. Ε, είναι λοιπόν θέματα πολύ σημαντικά τα οποία νομιμοποιούν τις δραστηριότητες σύμφωνα με την εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας διότι πρέπει να καλύπτουμε τα θέματα του χώρου της ε, δημοκρατίας, ελευθερίας και ασφαλείας για να μπορούν να συμμετέχουν και περισσότερο οι πολίτες σε αυτά τα πολύ ευρέστητα θέματα που δημιουργούν και διενέξεις. Ε, ε, όλοι υποκείμεθα σε πολλούς κινδύνους όπως η τρομοκρατία, το εμπόριο ανθρώπων και ε, ε, τα εγκλήματα είναι διασυνοριακά. Οι εγκληματίες εποφιλούνται των νέων τεχνολογιών και βλέπουμε και μία όλο και πιο έντονη δραστηριοποίηση διαφόρων ομάδων και γι' αυτό θα πρέπει να συμπληρώσουμε την εργασία των Εθνικών Κοινοβουλίων που είναι βασικά διότι το θέμα εσωτερικής ασφαλείας είναι δικαιοδοσία των κρατών μελών αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη εφαρμόζει τα θέματα τα οποία ε, έχουν ε, συμφωνηθεί και ε, υπάρχει μία στρατηγική Έχουμε δε ε, διαπιστώσει τέσσερις τομείς προτεραιότητος όπου μπορεί ε, να υπάρχει ε, συνεργασία για την τρομοκρατία, για το κυβερνοέγκλημα, για την ενίσχυση των εξωτερικών μας συνόρων και το πέμπτο είναι οι ανθρωπογενείς καταστροφές. Ε, είναι λοιπόν ένα πρόγραμμα το οποίο συμμερίζονται και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη για να προχωρήσουν τα επόμενα τέσσερα χρόνια και συνεργάζονται και επί καθημερινής βάσεως για την εφαρμογή αυτής της στρατηγικής. Ο ρόλος των οργανώσεων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως επίσης προχωρά και θα, θα συζητήσουμε για αυτές αργότερα σήμερα το απόγευμα και αύριο οι δυνατότητες αυτών των οργανώσεων μπορούν ε, να χρησιμοποιηθούν καλύτερα σε στενή συνεργασία και ο πρόεδρος θα παρουσιάσει ε, μία πρόταση για την αναθεώρηση και αναμόρφωση της Europort για να ε, προωθήσει την καταπολέμηση του εγκλήματος και θέλουμε επιπλέον η ΣΥΠΟΛ να γίνει μία οργάνωση η οποία θα μπορέσει να ενταχθεί καλύτερα στο πρόγραμμα εκπαίδευσης που Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να εφαρμόσει του, του χρόνου. Αλλά το πιο βασικό είναι η λογοδοσία, διότι αυτό μόνο νομιμοποιεί τους οργανισμούς αυτούς, αυξάνοντας την ε, ε, την ε, παρουσίαση και γι' αυτό θα πρέπει όλοι να δίνουμε όλο και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις οργανώσεις προς τα κοινοβούλια. Η Frontex είναι ένα καλό παράδειγμα για το πώς μπορεί να βελτιωθεί αυτή η οργάνωση διότι κάθε χρόνο παρουσιάζουμε μία έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη σειρά του μεταδίδει τις πληροφορίες αυτές. Βεβαίως υπάρχει νέα διακυβέρνηση του Σέγγεν και υπάρχει μία πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που ανέρχεται σε δύο εβδομάδες για τη βελτίωση της κατάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλες οι προτάσεις πρέπει να έχουν εγκριθεί ε, σύμφωνα με το άρθρο 87 της Συνθήκης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα γίνεται γίνεται η πρώτη έκθεση σχετικά με την ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα υιοθετηθεί τον Νοέμβριο για να κάνουμε έναν απολογισμό και να σχεδιάσουμε το μέλλον. Ε, έχουμε, έχουν όλοι οι οργανισμοί συμβάλει στην κατάρτιση της εκθέσεως αυτής και όλα τα θέματα συνεχίζουν ε, να υφίστανται, δεν είναι μεγάλη σημασία και πρέπει να δραστηριοποιηθούμε και στο μέλλον. Για το οργανωμένο έγκλημα η υπάρχει πρόοδος ε, σχετικά με τον έλεγχο ε, των διαβατηρίων για όσους εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, έχουμε και μία ε, μια οδηγία σχετικά με την ε, εμπορία ανθρώπων που τονίζει το θέμα αυτόν. Επιπλέον όμως ε, πρέπει να αυξήσουμε τις προσπάθειες για την καταπολέμηση σοβαρών εγκλημάτων να υπάρχουν αποτελεσματικές ομάδες που θα χρησιμοποιούνται πιο συχνά στο μέλλον και τα επιτεύγματά μας επέτρεψαν να καταρτήσουμε προενός μηνός ένα δίκτυο το οποίο επιτρέπει ε, να ε, εντοπίζουμε ορισμένους τρομοκάρατες οι οποίοι ε, χρηματοδοτούν την εγκληματικότητα και οι δράσεις ε, επίσης προχωρά κατά του κυβερνοεγκλήματος και ε, υπάρχει ένα κέντρο για το οποίο έχουν καταρτιστεί κατευθυντήριες γραμμές ε, και καταρτίζονται ομάδες για να ανταποκρίνονται στα προβλήματα μέσω των υπολογιστών. Όσον αφορά το διασυνοριακό έγκλημα, η πρόταση της Επιτροπής θα υποβληθεί ακολουθεί το Δεκέμβριο και η τελευταία προτεραιότητά μας ε, ε, η οποία προχωρά αλλά λιγότερο γρήγορα ε, αναφέρεται στην αξιολόγηση των κινδύνων σχετικά με την διαχείριση των καταστροφών και την αξιολόγηση των κινδύνων αλλά χρειάζεται εκεί μεγαλύτερη προσπάθεια για να προχωρήσουμε θα πρέπει να συνεχίσουμε συνεργάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα κράτη-μέλη περισσότερο και όπως είπα και στην αρχή για όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων που τώρα ενσωματώθηκαν στη συνθήκη της Λισαβόνας. Ολοκληρώνοντας λοιπόν θεωρούμε ότι τα εθνικά κοινοβούλια έχουν μεγάλη σημασία μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας και βλέπουμε ότι ακόμη και αν τα διάφορα θεσμικά όργανα πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες εξελίξεις προχωράμε καλά. Υπάρχει μία στρατηγική η οποία εξετάζεται και η σχετική έκθεση καταρτίζεται από την κυρία Μποσελίνο και ελπίζω ότι θα την ακούσουμε σύντομα. Ε, όσον αφορά την ασφάλεια και τα εσωτερικά κοινοβούλια δεν μπορεί να υπάρξει η ασφάλεια χωρίς ε, την δημοκρατική λογοθεσία και, ε, λογοδοσία και πρέπει να λάβουμε μέτρα για να μπορέσουμε να την ε, εφαρμόσουμε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Τώρα. Κυρία Θα ακούσουμε τον κύριο Ανταμραπάτσκι ο οποίος είναι αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Δίκησης της Δημοκρατίας Πολωνίας, πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής Εσωτερικής Ασφάλειας της ΚΟΖΗ, θα τοποθετηθεί εκ μέρους Πολωνικής Προεδρίας του Συμβουλίου και στη συνέχεια θα ακούσουμε άλλα δύο μέλη του Κοινοβουλίου, την κυρία Ρίτα Μπορσελίνου, που είναι η συγγήτρια ε, για την ε, στρατηγική ιστορική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον καθηγητή Τζουζέπε Κατάλμπη από ε, το Πανεπιστήμιο της Νάπολη. Κύριε Πρόεδρε, έλαβα αυτή την ε, πρόσκληση με μεγάλη ικανοποίηση για να συμμετάσχω σε αυτή την συνεδρίαση ε, η οποία θα εξετάσει την ε, στρατηγική εσωτερική ασφαλείας. Είναι μεγάλη τιμή ε, να μιλώ και να συζητώ με τόσο υψηλά ιστάμενους ομολόγους και ιδίως αφού έχω ασχοληθεί επί 20 χρόνια με την εσωτερική ασφάλεια στην Πολωνία. Ε, έχω αφιερωθεί ε, και διαπιστώσει τον αγώνα ε, κατά της εγκληματικότητας και υπέρ της εσωτερικής ασφαλείας και εδώ και 1,5 χρόνο η εσωτερική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως έχει εφαρμοστεί μέσω της νέας στρατηγικής ε, ε, διότι προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε απελές οι οποίες δεν αναφέρονται μόνο σε ενέργειες εντός των κρατών μελών αλλά και διασυνοριακά. Πρέπει όμως να αντιμετωπίσουμε όλα τα θέματα αυτά μαζί διότι δεν μπορούμε να ε, καταπολεμήσουμε καμία μορφή εγκλήματος χωρίς τη διεθνή συνεργασία και γι' αυτό βλέπουμε ότι τα μέτρα τα οποία χρησιμοποιούμε για να εφαρμόσουμε τις διατάξεις πρέπει να βασίζονται σε κοινέ αξίες όπως είναι ο ε, δημοκρατικό, το δημοκρατικό κράτος δικαίου και σαν εκπρόσωπος της αστυνομίας και των αρχών εφαρμογής της εσωτερικής ασφαλείας ε, σε διάφορα επίπεδα ε, θέλω να πω ότι θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι πολίτες θα είναι ασφαλείς και να ισοσκελίσουμε αυτό το στόχο με το σεβασμό των δημοκρατικών δικαιωμάτων. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει μία αναλογική αντιμετώπιση της ασφάλειας και οι δράσεις μας να είναι στοχευμένες. Πρέπει δηλαδή να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ένα επίπεδο ασφαλείας και ε, ότι αυτό αυτό θα γίνεται χωρίς να βλάπτουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η στρατηγική αυτή απαιτεί να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία πολιτών τρίτων χωρών και θα πρέπει και εκεί να βρεθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ της ανάγκης να ε, επεξεργαστούμε αυτά τα δικαιώματα συγχρόνως όμως ε, προστατεύοντάς τα. Ε, θα πρέπει λοιπόν γι' αυτό το λόγο να μπορέσουμε να προστατεύσουμε καλύτερα τους πολίτες και τα προσωπικά τους δεδομένα ότι ε, τώρα όταν συγκεντρώνουμε και ε, αποθηκεύουμε ε, στοιχεία θα πρέπει να βασιζόμαστε στην αρχή της νομιμότητος και της αναλογικότητος διότι τα στοιχεία αυτά είναι εμπιστευτικά και η εποπτεία από ανεξάρτητα όργανα θα πρέπει να είναι ισοσκελισμένη. Δηλαδή ε, πρέπει απλούστατα να χρησιμοποιούμε τα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά θα πρέπει να τα προστατεύουμε συγχρόνως και θα πρέπει να προφυλάξουμε καλύτερα καλύτερα για όλους τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ενώσεως ιδίως ε, αυτών οι οποίοι έχουν ε, μειωμένες δυνατότητες να παρακολουθήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία πρέπει να γνωρίζουν τι συμβαίνει πώς ε, διαχειριζόμαστε τα προσωπικά τους δεδομένα ότι τα δεδομένα αυτά ελέγχονται και προστατεύονται κατά την επεξεργασία αυτή λοιπόν η ισορροπία μεταξύ της προστασίας των δεδομένων και των ε, αναγκών ε, για την ε, εφαρμογή μιας δημόσιας στρατηγικής αντιμετωπίζουμε μία πρόκληση και αυτή είναι η πρόκληση και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για τα Εθνικά Κοινοβούλια και πρέπει να καταφέρουμε τα στοιχεία αυτά να ε, ε, καταγράφονται, να αποθηκεύονται και να επεξεργάζονται αλλά ε, μέσα σε ένα σωστό πλαίσιο ιδίως ε, όταν πρόκειται για επιχειρησιακούς ελέγχους στα πλαίσια των οποίων συγκεντρώνονται τα στοιχεία αυτά πρέπει να υπάρχουν ε, και να γίνονται σοβαστές οι προθεσμίες ε, του χρόνου διατηρήσεως των στοιχείων αυτών και μπορεί και τα εθνικά κοινοβούλια να προβούν σε επερωτήσεις ή να μας υποδείξουν πώς πώς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε περαιτέρω τα στοιχεία αυτά. Κατά την ε, Πολωνική Προεδρία το τμήμα μου ασχολείται με την πρόκληση της εσωτερικής ασφαλείας. Είναι μία μόνιμη επιτροπή η οποία εφαρμόζει μακροπρόθεσμα προγράμματα που ασχολούνται με τομείς απειλών που έχουν καθοριστεί. Υπάρχουν συγκεκριμένοι ε, στόχοι και στρατηγικά προγράμματα για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ε, προκλήσεις και προσμονές. Ε, επίσης πρέπει να φροντίσουμε όταν εφαρμόζουμε την στρατηγική της εσωτερικής ασφαλείας να διατηρήσουμε την ασφάλεια και, ε, και τα δικαιώματα των πολιτών. Γι' αυτό και η Πολωνία προσπαθεί στον τομέα της στρατηγικής της εσωτερικής ασφαλείας ε, να ε, συνδυάσει ε, το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και γι' αυτό υπάρχει και το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ και τώρα δίνουμε το λόγο μας εις την εισηγήτρια για το θέμα, την κυρία Μπορσελίνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, πέρασε ένα έτος από την τελευταία συναντήσή μας και δύο χρόνια από τη θέση σε σχέση τη συνθήκη τη Λισαβόνα ε, και ε, χάρτη των Μελιωδών Δικαιωμάτων. Ε, Όμω η νέα συνθήκη αποτέλεσε ένα πραγματικό ποιοτικό άλμα ιδίω για τι πολιτικέ που συνδέονται με την μεταμόρφωση τη Ένωση, σε ένα χώρο δικαιοσύνη, ελευθερία και ασφάλεια. Αν πριν από τη Λισαβόνα η Ένωση έπρεπε να ευνοήσει κυρίω τη συνεργασία μεταξύ των δικήσεων και να περιοριστεί στον προσδιορισμό καθορισμό των ελάχιστων κοινών κανόνων όπως πολιτική ασύλου κατόπιν αυτού είναι οι ίδιες συνθήκες που μας, επι... που μας επιβάλλουν να οικοδομήσουμε μια κοινή πολιτική σε ό,τι αφορά την προστασία των συνόρων, μεταναστευτική πολιτική και ασύλου. Και στο θέμα της εσωτερικής ασφάλειας μας ζητείται να ξεπεράσουμε τις εθνικές στρατηγικές και να δράσουμε και σε εθνικό επίπεδο με μια ευρωπαϊκή προοπτική. Σε αυτή την προοπτική, σύμφωνα με το άρθρο 2 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωση και τα Εθνικά Κοινοβούλια πρέπει να συνεισφέρουν στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα χωρίς ε, φυσικά να εγκαταλείψουν ε, την ε, διμερή προνομιούχο σχέση με τις αντίστοιχες κυβερνήσεις. Στους κύριους αυτούς μόνο αν επιβληθεί μια ευρωπαϊκή προοπτική μπορούμε να ξεπεράσουμε τις προκλήσεις που επιφέρει η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης τόσο οικονομικό τομέα, στον οικονομικό τομέα όσο και στον τομέα του ελέγχου των συνόρων και των μετασταυτικών ροών. Στον οικονομικό τομέα τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακαλύψε ότι δεν είχε αναπτύξει επαρκώς ε, εργαλεία βέα αλληλεγγύης που θα έπρεπε να συνοδεύσουν ε, τη δημιουργία του ενιαίου και τώρα προσπαθεί ε, να επιδιορθώσει την κατάσταση. Εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα το ίδιο να γίνει για τις πολιτικές που σχετίζονται με το χώρο ελευθερίας δικαιοσύνης και ασφάλειας όπου επικινδύνος. Ε, τελευταία βλέπουμε να πολλαπλασιάζονται ε, τα μηνύματα, τα σημάδια αμοιβαία δυσπιστίας απέναντι στα κράτη-μέλη, παραδείγματος χάρη σε ό,τι αφορά την επανεισαγωγή των ελέγχων στα σύνορα. Αυτές πρωτοβουλίες αιτιολογούνται με την επίκληση του κινδύνου που διατρέχουν οι πολίτε ενώ τα άλλα κράτη-μέλη θεωρείται ότι δεν προσφέρουν πλέον τις ίδιες εγγύσει για να διατηρηθεί η ελευθερία της κυκλοφορίας, που για το χώρο δικαιοσύνη ελευθερίας και ασφάλειας είναι αυτό που είναι το ευρώ για την εσωτερική μα αγορά. Έτσι λοιπόν, κατά την άποψή μου, αυτά τα δύο μόνο συμβαδίζουν, δείχνοντας μεγαλύτερη αλληλεγγύη και κοινή δέσμευση και σοβαρότητα και όχι ε, καταφεύγοντας σε κάποιες εφήμερες ε, λαϊκιστικές ε, ε, δράσεις. Η συνθήκη η ίδια στο άρθρο 80 μάλιστα μας επιβάλλει αυτή την αλληλεγγύη που δεν είναι μόνο οικονομική. Και αυτό προκύπτει τουλάχιστον ε, εν μέρη από του στόχου που καθορίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο πρόγραμμα τη Στοκόλμη και από τι ε, στρατηγικέ που υιοθετήθηκαν, ε, όπω η στρατηγική εσωτερική ασφάλειας που υιοθετήθηκε πέρσι. Στην προοπτική αυτή και στην προοπτική τη πιστή συνεργασία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε, παραδείγματο χάρη, Βουλγαρία και Ρουμανία να αρχίσουν να αναπτύσσουν ε, ε, τις λειτουργίες που σχετίζονται με ε, το χώρο Σένγκεν. Αυτές οι χώρες ε, είχαν ουσιαστικά σεβαστεί τις απαιτήσει. έτσι λοιπόν δεν μου φαίνεται ότι τώρα είναι ορθορισμένες κυβερνήσεις να επικαλούνται νέες συνθήκες αν και φυσικά κάθε παίκτη του χώρου Σένγκεν επιφέρει κάποιους κινδύνους αλλά θα πρέπει να προσφέρουμε τη δυνατότητα συμμετοχή σε αυτέ τι χώρε. Αν θέλουμε να καταστήσουμε πιο σοβαρού αυτού του ελέγχου και τι αμοιβέ αξιολογήσει, τόσο το Κοινοβούλιο όσο και η Κομισιόν είναι διαθέσιμα έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την ε, ε, ασφάλεια όλων των πολιτών και όλων της επικράτειας και όχι μόνο του κάθε κράτους. Τώρα να επανέλθουμε στο θέμα της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας. Ανυπομονούμε τώρα να λάβουμε από την Κομισιόν την πρώτη ετήσια έκθεση εφαρμογής της και θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο για αυτή τη διήμερη συζήτηση να είχαμε λάβει την έκθεση και Εύχομαι το επόμενο έτος Καθώ ελπίζω ότι θα ενωθεί αυτή η κοινοβουλευτική πρωτοβουλία, δεύτερη ετήσια έκθεση να είναι στη διάθεσή μα εγκαίρω και επίσης ελπίζω η Επιτροπή εσωτερική ασφάλεια η ΚΟΖΗ, να μα στείλει μια έκθεση πιο λεπτομερή σε σχέση με αυτή που μας έστειλε φέτο και που θα βρείτε στου φακέλου. σα. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι η σημερινή ανταλλαγή πληροφοριών ε, σε διοργανικό επίπεδο δεν είναι ικανοποιητική όπως προκύπτει και από τα ψηφίσματα που θετήθηκαν ε, πρόσφατα στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕΣ ό,τι αφορά το θέμα της, ε, των πληροφοριών για θέματα όπως η καταπολέμηση τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Αναφέρομαι στην εκθέση Ελφάνου παραδείγματος χάρη η σύγχυση αυτή είναι ακόμα μεγαλύτερα αν βλέπουμε ότι στα άρθρα 70 και 71 σε ό,τι αφορά ε, την ενημέρωση των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η συνθήκη είναι κάπως μετριόφρον. Λεχθέντος ε, αυτού, οι συζητήσεις μας αυτό το διήμερο ελπίζω να βρήθουν ενδιαφέροντων ιδεών που θα ακούσουμε και για τους, ε, τον έλεγχο των οργανισμών Frontex, Europol και Eurojust επίσης. Εμείς ε, για να καλύψουμε το επίσημο κενό πληροφοριών ζητήσαμε την οργάνωση αυτής της συζήτησης. Ελπίζω να ενδιαφέρει και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Πρόκειται και για μία μελέτη για το ρόλο των ε, ευρωπαϊκών οργανισμών για το ρόλο που διαδραματίζουν όταν θέτουν σε εφαρμογή την στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας. Προσωπικά, αν και εκτιμώ τη σοβαρότητα των ενδείξεων και τη μεθοδολογία που προτείνονται, θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο επόμενο πολιτικό κύκλο ασφαλεία που θα πρέπει να ξεκινήσει το 2013 να προσδιοριστεί χωρί ε, να υπάρχει ε, μία διάρθρωση και μία συμμετοχή Εθνικών Κοινοβουλίων ε, και Ευρωκοινοβουλίου. αυτή η μελέτη εν μερή απαντά σε ορισμένες κριτικές ε, που έγιναν στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς ε, όταν παρεμβαίνουν ε, χωρίς να χρειάζεται σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές. Νομίζω ότι τις κριτικές πρέπει να ληφθούν υπόψη και στην περίπτωση αυτή η συνθήκη προβλέπει τη συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων στον έλεγχο της Ευρωπόλ και της Eurojust, αλλά δεν βλέπω γιατί αυτός ο έλεγχος δεν θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλους οργανισμούς ε, που έχουν παρόμοια καθήκοντα όπως η Frontex. Παραδείγματο χάρη, καθώς βλέπουμε ότι προοδευτικά δημιουργείται μια σειρά οργανισμών ε, ε, όπου οι εθνικές διοικήσεις εκπροσωπούνται, όμως δεν υπάρχει πραγματική κοινοβουλευτική ευθύνη. Και τέλος, μια μελέτη που ε, να συγκρίνει πώς έχει η κατάσταση της πρόσβασης των Εθνικών Κοινοβουλίων σε απόρριτες πληροφορίες. Πρόκειται για μια πολύ χρήσιμη μελέτη, γιατί όπως εξήγησα και στα έγγραφα εργασία μου, είναι αναπόφευκτο όταν πρόκειται για θέματα ασφάλειας, είτε εσωτερική είτε εξωτερικής. Κάποιες πληροφορίες πρέπει να είναι απόρριτες ε, για να μην τεθεί σε κίνδυνο τα συμφέροντα των κρατών μελών και της Ένωσης. Όμως αυτό δεν πρέπει να γίνει καταφύγιο για να παρεμποδίζεται η πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές από τους εκπροσώπους ε, των ε, πολιτών. Και υπάρχει απουσία κάποιων κανόνων σε ό,τι αφορά τη διαβάθμιση και τον αποχαρακτηρισμό των εγγράφων. Και οποιοδήποτε υπάλληλος ε, ε, ουσιαστικά είτε σε εθνικό είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο τελικά έχει υπερβολική εξουσία για να αποφασίσει αν θα επιτρέψει την πρόσβαση ή όχι στα ίδια τα έγγραφα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η κατάσταση είναι αν μη τι άλλο μπερδεμένη θολή και έτσι λοιπόν θα ήθελα με την έκθεση Κάσμα να βρούμε και μία νομική λύση πιο κατάλληλη σε σχέση και με αυτό που λέγω τη συνθήκη και αποφασίστηκαν και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν ε, θα βρείτε ε, στα έγγραφά σας ε, το σχέδιο εκθεσινού γιατί σκοπεύω να του προσθέσω κάποια στοιχεία κατόπιν των συζητήσεων με τους σκιώδες συζητητές και κατόπιν διαβουλεύσεων με την Κομισιόν και με το Συμβούλιο. Τελευταία παρατήρηση. Μέχρι τα τέλη του έτους θα προσπαθούσουμε να οργανώσουμε τη συνάντηση του επόμενου έτους ε, για τη στρατηγική εσωτερική ασφάλεια, έτσι ώστε να μπορούσουμε καλύτερα να οργανωθούμε και να προετοιμάσουμε ίσως και εθνικέ εκθέσεις που θα μας επιτρέψουν να έχουμε μια καλύτερη εικόνα της κατάστασης. Και φυσικά εδώ τα αφήνω στα χέρια της Προεδρίας να εξάγει τα σχετικά συμπεράσματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Μπορσαλίνο. Τώρα ένας τελευταίος γύρος σε αυτό το πρώτο μέρος των εναρκτηρίων δηλώσεων ο καθηγητής Τζουζέπε Κατάλντι που θα μας κάνει έτσι την, θα μας εκφράσει την άποψη του ακαδημαϊκού εμπειρογνώμονος της εξισορρόπησης μεταξύ ασφαλείας και θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ορίστε καθηγητά μου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ παρουσίασα μία σύντομη ομιλία στα αγγλικά, αλλά θέλω στη γλώσσα μου να ευχαριστήσω εσάς και τους οργανωτές αυτή της συνάντηση επειδή μου, δώσετε, μου δίνετε ε, τη δυνατότητα να εκφράσω και μία ακαδημαϊκή άποψη, όπως είπατε κι εσείς. Και ε, φυσικά σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να επιτελέσω αυτό το καθήκον και ε, προσωπικά, αλλά και ως αντιπρίτανης. Θα προσπαθήσω τώρα να σας μιλήσω κυρίως για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σύμφωνα με τη χάρτα, ελευθερία, δικαιοσύνη, ασφάλεια του ατόμου. Δύο χρόνια μετά την θέση ενισχύ της Συνθήκης Λισαβόνας και της Χάρτας, φαίνεται ότι δεν έχουν γίνει ακόμη αρκετά νομοθετικά. Νομοθετικός και δίνεται όλη η προσοχή στη διακυβερνητική μέθοδο και μόνο στην ασφάλεια. Εδώ θα προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε την ομολογία, δηλαδή το δόγμα του περιθωρίου ερμηνείας που δίνει το δικαστήριο και που δεν έχει τύχει εκμετάλλευσης μέχρι τώρα για να την αντιμετώπιση του λεπτού θέματος της εξισορρόπησης της εσωτερικής ασφαλείας με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το περιθώριο αυτό θα μπορούσε να υποκατασταθεί από θεωρία σε πράξη. Θα μπορούσε κανείς να συγκρίνει από τη μια τα δικαστήρια με την άλλη τα κοινοβούλια. και τα δύο είδη οργάνων έχουν δικαιώματα και υπευθυνότητε. Αλλά η δημιουργία νέων δικαιοδοσιών πρέπει παράλληλα να εξισορροπηθεί με την ανάγκη της κοινοβουλευτικής εποπτείας όπως προβλέπει η συνθήκη της Λισαβόνας αλλά που δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί ούτε στρατηγικά, ούτε νομοθετικά, ούτε λειτουργικά. Βέβαια υπάρχουν εδώ δυσκολίες. Θα αναφέρω μερικές από αυτές. Το πρόβλημα των υπηκών τρίτων χωρών σε αυτόν τον χώρο ελευθερίας, ασφαλείας και δικαιοσύνης δεν πρέπει οι πολίτες αυτοί, δηλαδή τρίτων χωρών, να πληρώνουν την ύφη για τη δημιουργία αυτού του χώρου. Στις αρχές του φιλόδοξου αυτού οράματος, το θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων είχε τεθεί και δεν είναι το μόνο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Είναι και θέμα ανθρωπισμού και πολιτισμού, πεπολιτισμένης συμπεριφοράς. Δεν θα είχε νόημα να οικοδομηθεί εδώ ένα ευρωπαϊκό φρούριο που να τους αποκλείει. Έπειτα υπάρχει και η συνεργασία, διότι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, παράλληλη εφαρμογή στρατηγικών ασφαλείας είναι δύσκολο πράγμα ως προς τη συνεργασία με τρίτες χώρες και τις υπηρεσίες τους. γιατί αυτές οι υπηρεσίες τρίτων χωρών δεν έχουν πάντοτε τα ίδια ενδιαφέροντα με τις Ένωσης. Δεν αρκεί λοιπόν να σταυρώσουμε τα χέρια, πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω για να εφαρμόζονται τέτοιου είδους συμφωνίες με τρίτες χώρες πραγματικά. Πρέπει να προασπιζόμαστε πάντοτε τα ελάχιστά μας κριτήρια. Ξέρετε την απόφαση Γιουσούφ Ελκάντη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που έδειξε καθαρά ότι το επίπεδο προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων που εξετάζει και ο ΙΕ ακόμη για την καταδίκη τρομοκρατών δεν μπορεί να παραβιάζει το κοινοτικό κεκτημένο. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα τώρα να σας υπενθυμίσω ποια είναι Ποιο είναι αυτό το δόγμα της, ε, του περιθωρίου ερμηνείας. Γενικά η έκφραση αυτή αναφέρεται στις δυνατότητες που έχει το δικαστήριο του Στρασβούργου, που διαθέτει το δικαστήριο του Στρασβούργου στις εθνικές αρχές για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εδώ οι λέξεις κλειδιά είναι γνωστές. Επικορικό και επιτήρηση, εποπτεία. Το δικαστήριο του Στρασβούργου είναι σε συνεχή επαφή με τις εθνικές αρχές και είναι σε θέση, που είναι σε θέση καλύτερα από ότι εκείνο να ερμηνεύσει την ομολογία. Αλλά οποιαδήποτε παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι απαράδεκτη γιατί πρέπει πάντοτε να σεβόμαστε ορισμένα ελάχιστα κριτήρια. Η σχέση μεταξύ ευρωπαϊκών νομοθετικών σωμάτων του Ευρωπαϊκού δηλαδή Κοινοβουλίου και των Εθνικών και των υπηρεσιών εσωτερικής ασφαλείας πρέπει να βασίζονται στα εργαλεία που έχουν δοκιμαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έτσι ώστε η συνεργασία εθνικών και υπερεθνικών επιπέδων να είναι η καλύτερη. Θα έπρεπε να εξεταστεί η δυνατότητα εκμετάλλευσης περαιτέρω αυτού του δόγματος. Παραδείγματο χάρη όταν ένα κράτος ερμηνεύει κάποια απειλή που βλέπει. Βέβαια πρέπει να είναι περιορισμένο αυτό το περιθώριο, περιορισμένο. Γιατί θα υπάρχει και η επιτήρηση από το διεθνή παράγοντα, από τον υπερεθνικό μάλλον παράγοντα για να μην ξεπερνούνται τα πλαίσια και όρια της νομιμότητας. Οι παράμετροι που πρέπει να εφαρμόζονται είναι γνωστές. Προσβασιμότητα, ύπαρξη μη θεμητού στόχου και αναλογικό της ε, η χρήση λοιπόν αυτού του περιθωρίου θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι ένα συγκεκριμένο εργαλείο στα χέρια όλων όσων θέλουν να σεβαστούν το άρθρο 7.2 της Ιθήκης Στοκόλμης για το σεβασμό των ανθρωπίνων και θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό επίσης διότι υπάρχουν ακόμη, ακόμη λέγω, προβλήματα ως προς προς τον τρόπο με τον οποίο οι υπηρεσίες αυτές αντιδρούν. Σας υπενθυμίζω το Bundesverfassungsgericht του Ιουνίου 2009 που θεωρεί τη συνθήκη της Λισαβόνας μεν συμβατή με το γερμανικό σύνταγμα αλλά σπέβδει να κάνει μια στενή ερμηνεία της ε, ως προς τον ιδιωτικό χώρο και τα δικαιώματα των πολιτών. Αυτό είναι σύμπτωμα μιας θεμητής ανησυχίας που μπορεί να δημιουργεί στις εθνικές αρχές η συνθήκη της Λισαβόνος. Υπάρχει λοιπόν ένα πρόβλημα εδώ δημοκρατικής λογοδοσίας για να οικοδομηθεί αυτός ο χώρος ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφαλείας και δεν πρόκειται εδώ για απλό ευσεβή πόδο αλλά για νομική υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 10 και το άρθρο 2 της συνθήκης της Λισαβόνας. Έτσι καταλήγω. Πρέπει να λυθεί αυτό το θέμα της λογοδοσίας και της, και της ευθύνης και χρήσιμότερο εργαλείο από όλα θα ήταν η χρήση αυτού του περιθωρίου ερμηνείας που ανέπτυξε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά Κατάλτη. Τώρα, όπως είπαμε, έχουμε περίπου 40-45 λεπτά στη διάθεσή μας για τη συζήτηση. Θα πρότεινα να δώσουμε το λόγο σε δύο μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων και κατόπιν σε ένα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έτσι ώστε να δίνουμε το λόγο με τη σειρά. Θα ξεκινήσουμε από τον Λόρδο Δαβιτχανέ, από τον οίκο των Λόρδων, του Ηνωμένου Βασιλείου. Παρακαλώ. Ο Λόρδος Χανέη. Ευχαριστώ για το λόγο, Πρόεδρε. Θα ήθελα να δράξω την ευκαιρία να σχολιάσω την έκθεση της ε, Επιτροπής μου για την στρατηγική ασφάλειας. Ε, ο πυρήνας της εκθέσης αυτής ήταν ότι η εσωτερική ασφάλεια, ενώ είναι εθνική ευθύνη, ούτε ξεκινά ούτε τελειώνει στα εθνικά σύνορα. Και αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται συλλογική δράση αλλά και εθνική δράση. Και το δεύτερο σημείο που τονίσαμε είναι ότι πιστεύουμε ότι η Κομισιόν έχει εντοπίσει τις πέντε προτεραιότητες κατά πολέμηση τρομοκρατίας, ε, ε κυβερνοχώρος, οργανωμένο έγκλημα, έλεγχος των συνόρων ε, και αντιμετώπιση καταστροφών. Είναι σωστές αυτές οι προτεραιότητες και σωστά επικεντρώνεται σε αυτές. Τα κύρια συμπεράσματα ήταν ότι η εσωτερική ασφάλεια πρέπει να συμβαδίζει με την εξωτερική ασφάλεια και η Κομισιόν πρέπει να κάνει περισσότερα από όσα στο παρελθόν ε, για να συμβαδίζουν αυτά τα δύο και για να υπάρχει καλύτερο συντονισμός. Δεύτερον, Υποστηρίζουμε αν θερμά την αναγκή για την αναγνώριση της νομοθεσίας ε, για τους καταλόγους ονομάτων επιβατών, PNR, και νομίζουμε ότι θα είναι πιο αποτελεσματική αν εφαρμοζόταν ε, και σε πτήσει εντό Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο σε πτήσει που έρχονται εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίση ε, μα προβλημάτισε που η Κομισιόν δεν αναφερόταν ε, στην αντιμετώπιση των καταστροφών στο ρόλο του στρατού. Βλέπουμε, παραδείγματο χάρη, στην περίπτωση τη Ιαπωνία, όπου είχαμε το τσουνάμι, πω σε μια πραγματικά μείζωνα καταστροφή είναι ο ρόλος του στρατού κρίσιμος ε, στα αρχικά στάδια. Έτσι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να σκεφτεί πώς θα συντονίσει αυτή τη δραστηριότητα. Και το τελικό συμπέρασμα ήταν, και φοβάμαι να πω ότι εξακολουθούμε να, πιστεύω, να πιστεύουμε ότι υπάρχουν υπερβολικά πολλοί φορεί στο Συμβούλιο που, που ασχολούνται με τα θέματα αυτά και χρειάζεται κάποιο εξορθολογισμό στα επόμενα χρόνια. Και αυτό χωρίς να εκφράζουμε ε, ουσιαστικά λήψη σεβασμού για τον Υπουργό Ραπάτση και εμείς ε, ότι υπήρχε δυνατότητα ε, να, η Προεδρία της Κόζη να μην είναι εκ αλλά να έχει επιλεχθεί κάποιος πρόεδρος από την Επιτροπή για μία περίοδο δύο χρονών όπως γίνεται στην περίπτωση Frontex και Europol προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη συνέχιση. Όμω, ε, η κύρια έμφαση μα ε, ήταν στον κυβερνοχώρο. Αποτελεί αυτό σε ένα νέο τομέα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και καθημερινά καθίσταται μεγαλύτερη απειλή για την εφημερία και την ασφαλειά μας. Ε, ήδη όταν ε, συντάξαμε την εκθεσή μας ε, είχαμε κάποια παραδείγματα σε σχέση με την επίθεση που δέχονται οι θεσμοί, δηλαδή και η υπηρεσία εξωτερικής δράσης και το σύστημα εμπορίας εκπομπών δέχτηκαν επίθεση και δυστυχώς δεν τα πήγαν και πολύ καλά στη διαχείριση γιατί δεν είχαν τον κατάλληλο εξοπλισμό και πιστεύουμε ότι το κράτη-μέλη θα πρέπει να ενδυναμώνουν την ικανότητα των θεσμών ορισμένα κρατημέλη έχουν επαρκεί γνώσει και δεξιότητε στον τομέα αυτό. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να βοηθήσουν του θεσμού να οικοδομήσουν την αμυνά του, έτσι ώστε να μην ε, έχουμε ε, ενδημικό φαινόμενο. Συμφωνούμε με την Κομισιόν ότι πρέπει να υπάρχει ένα κέντρο για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και ελπίζουμε ότι η Επίτροπο όταν θα παρουσιάσει προτάσει ε, θα αναθέσει αυτό το καθήκον στη Europol. Γιατί εμεί θεωρούμε ότι αυτή είναι η κατάλληλη υπηρεσία να το αναλάβει. Και Πρέπει να πω ότι διαφωνούμε με τη δική μας κυβέρνηση που πιστεύει ότι όλα όσα μπορούν ε, να γίνουν, ε, δηλαδή η σύσταση ενός τέτοιου κέντρου για τα πολέμηση του εγκλήματος στο κυβερνοχώρο με τους υφιστάμενους πόρους, κάτι τέτοιο εμείς δεν θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα αξιόπιστο. Αυτή την ε, έκθεση ήθελα να σας παρουσιάσω, τη σύνοψη την έχετε στα έγγραφα για αυτή τη συνεδρίαση. Ελπίζω όλοι να ρίξουν και μια ματιά στο σύνολο της έκθεσης και να σας πω ότι πραγματικά πρόκειται για ψήφο εμπιστοσύνη ε, ο τρόπο ε, με τον οποίο παρουσίασε τα καθήκοντά τη η Επίτροπο. Μάλιστα, ευχαριστούμε. Τώρα ο κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέρη από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι είναι πολύ μεγάλη η τιμή να συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία ως εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινοβουλίων και βέβαια έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία να βρισκόμαστε εδώ ενώπιον τόσο σημαντικών προσωπικότητων του ευρωπαϊκού γίγνεσθε. Όμως, για να έχει αξία και νόημα η διαδικασία του ελέγχου που ασκούμε στα πλαίσια αυτής της διακοινοβουλευτικής σύσκεψης, θα πρέπει πρώτον να γνωρίζαμε τι απέγιναν οι επισημάνσεις, οι υποδείξεις και οι υπογραμμίσεις που είχαμε κάνει πριν από ένα χρόνο μέσα σε αυτή την αίθουσα στα πλαίσια ακριβώς της ίδιας διαδικασίας. Δηλαδή, ποιας υποδοχής έτυχαν οι υποδείξεις που είχαμε κάνει, ο έλεγχος, σε πάση περιπτώσει, που είχαμε ασκήσει στα συγκεκριμένα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μία δεύτερη σκέψη ήθελα να πω. Ακούγοντας τους προλαλήσαντες, αυτούς οι οποίοι πολύ ορθά έθεσαν τα θέματα από την πλευρά των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρώ και πρέπει να το επισημάνω ότι έχουμε κυρίως υποχρέωση σε αυτές τις κρίσιμες ώρες που ζούμε όλοι μας και κυρίως οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου να αντιληφθούμε ότι ενδεχομένως θα πρέπει να δώσουμε πολύ μεγαλύτερη σημασία στην πολιτική και στη δημοκρατία παρά στις απόψεις κάποιων τεχνοκρατών οι οποίοι παραγνωρίζουν το γεγονός ότι η διαμόρφωση στρατηγικών εσωτερικής ασφάλειας όπως και η διαμόρφωση πολιτικών επάνω σε συγκεκριμένα θέματα που έχουν να κάνουν με τη διαμόρφωση του ενιαίου χώρου ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας έχουν αξία μόνο όταν αναφέρονται πρώτον σε δημοκρατίες, δηλαδή όταν αναπτύσσονται στα πλαίσια δημοκρατιών, δημοκρατικών δηλαδή καθεστώτων και δεύτερον όταν αποτελούν εκδηλώσεις πολιτικής, πολιτικής με πι κεφαλαίο. Γιατί δυστυχώς ήδη η ιστορία φοβούμε ότι έχει αλλάξει κήτη και εκεί που όλοι περιμέναμε αυτό το ευρωπαϊκό όραμα να φτάσει στην ολοκλήρωσή του φοβούμε μήπως οι αγορές δεν έχουν πει ακόμα τον τελικό τους λόγο γιατί από ό,τι φαίνεται οι δημοκρατίες και οι πολιτικές υποχωρούν μπροστά στην άσκηση των οικονομικών άτυπων διαδικασιών οι οποίες εκπορεύονται από τις λεγόμενες αγορές. Και προς αυτή βεβαίως την κατεύθυνση θα πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας γιατί έχουν σχέση και με τη, στρα... στρατηγική που πρέπει να διαμορφώνουμε για, τις για την εσωτερική ασφάλεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα... Ευχαριστώ. Τώρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η κυρία Τζούντιτ Σαρζεντίνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι ακούγοντας ε, τους ε, συναδέλφους αλλά και στους φιλοξενούμενους μας ε, δεν κατάλαβα τι σκέπτονται ότι αποτελεί το βασικό θέμα της εσωτερικής στρατηγικής διότι άκουσα για τους υπηκόους τρίτων χωρών που ανέφερε ο καθηγητής οι οποίοι ίσως ε, υποφέρουν ε, και ε, δεν εποφελούνται της στρατηγικής μας και βεβαίως θέλουμε να συνεργαστούμε στενά για να μπορέσουμε να καταρτήσουμε αυτό το χώρο εσωτερικής στρατηγικής να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερες διατάξεις όπως άλλωστε και μία ανάλυση της ε, ε, Europol σχετικά με τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και θα θέλαμε να ακούσουμε και την άποψη του Συμβουλίου διότι παραδείγματο χάρη όσον αφορά την ε, λαθρομετανάστευση η οποία αποτελεί πρόβλημα ή υπάρχει θέμα ασφαλείας υπάρχει ένα πρόβλημα ασφαλείας τα εθνικά κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν συμφωνούν σχετικά με ε, αυτά τα οποία παρουσιάζει η ανάλυση της ε, Europol και διαμορφώνουν ή διαγνώμη. Θα ήθελα όμως να ξέρω τι γίνεται στην πραγματικότητα και ποια είναι η έκβαση των αποφάσεων και αν αυτή θα είναι χρήσιμη. Ε, Διότι επιπλέον το θέμα αυτό συζητιέται και σε άλλα θέματα σχετικά με τα πλαστά τα εμπορεύματα, τα πλαστά φάρμακα ε, υπάρχουν διάφοροι τομείς διότι ενδεχομένως στην Ευρώπη δεν έχετε μεγάλο ποσοστό των φαρμάκων τα οποία κατασκευάζονται ε, σε τρίτες χώρες ε, και υπάρχει και ένα θέμα εργατικού δυναμικού αλλά το θέμα είναι πώς μπορούμε να διακρίνουμε τι είναι ασφαλές από αυτό το οποίο δεν είναι. Με συγχωρείτε. Αλλά θα υπάρχει θα υπάρξει και δεύτερος γύρος. Θα ακούσουμε ένα δεύτερο γύρο ερωτήσεων από Ευρωβουλευτή και Εθνικό Εκπρόσωπο και μετά θα γίνει ε, μία, ε, ένας γύρος απαντήσεων. Αλλά τώρα θέλω να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο ε, του Γερμανικού Κοινοβουλίου, του Bundestag Ευχαριστώ. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μια στρατηγική εσωτερικής ασφαλείας ε, διαφυλάσσοντας τα θεμελιώδη δικαιώματα και καθιερώνοντας τη δημοκρατική λογοδοσία και έχω μια ερώτηση σχετικά με, ε, που απευθύνεται στην κυρία Μάλστρομ για τα PNR. Αντιλαμβάνουμε ότι θα καταλήξει η συμφωνία τον Νοέμβριο και προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασκεδάσει τις αμφιβολίες και επιφυλάξεις που έχουν διατυπώσει οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών ε, τι πρόκειται να γίνει στο μέλλον διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 394 οι υπάλληλοι ε, στις Ηνωμένε Πολιτείες ε, υπάρχουν αποφάσεις σχετικά με 394 ε, περιπτώσεις που δεν θεωρήθηκαν ότι μπορούσαν να γίνουν αποδεκτές. Επίσης ε, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το τελευταίο τρίμηνο ε, πρόκειται να υπάρχει συνεργασία με την Τουρκία. Τι εννοείται στο θέμα αυτό διότι υπάρχει ένα ένα θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τη χώρα αυτή. Και τέλος μία ερώτηση στον καθηγητή Κατάλτη, ο οποίος μίλησε για την υποχρέωση της δημοκρατικής λογοδοσίας και αυτό αναφέρεται και στους οργανισμούς Ευρωπαϊκής Ενώσεως, στην Frontex, την Europol κτλ. Αντιλαμβάνουμε ότι έγινε μία μελέτη στο, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με το πρόβλημα του δημοκρατικού ελέγχου. Λοιπόν, τι γίνεται με τον δημοκρατικό ή μη δημοκρατικό έλεγχο αυτών των οργανισμών και πώς θα αντιμετωπιστεί στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Μπούμπλαντ από το Τσεχικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Έχω ένα σχόλιο σε ό,τι φορά την παρέμβαση της κυρίας Μπορσελίνου αναφέρθηκε σε ορισμένα προβλήματα με ε, το βαθμό της διαβάθμισης ε, των εγγράφων ε, και τον αποχαρακτηρισμό τους. Είναι ένα θέμα που το συζητάμε πολύ συχνά και αυτό το πρόβλημα ουσιαστικά καθίσταται εμπόδιο στο να επικοινωνήσουν μεταξύ τους οι αστυνομίες των διάφορων κρατών μελών. Εγώ πιστεύω ότι θα ήταν καλό να υιοθετήσουμε κάποιους κανόνες που θα μπορούσαν να είναι αντίστοιχοι με τους κανόνες που ισχύουν στο ΝΑΤΟ. Και κατόπιν να θεσπίσουμε την αρχή αυτός που έχει δημιουργήσει την πληροφορία να μπορεί να τη διαβαθμίσει γιατί αυτός ξέρει καλύτερα ε, ποιο πρέπει να είναι το επίπεδο της διαβάθμισης. Οι λοιποί θα πρέπει να σεβαστούν τη διαβάθμιση αυτή. Και Επίσης, ε, για την πρόσβαση στις πληροφορίες ε, πρέπει την πρόσβαση να την χορηγεί επίσης αυτός ε, που δημιουργεί την πληροφορία. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε ένα εσωτερικό σύστημα. Κατόπιν μπορούμε να θέσουμε το ερώτημα του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Το κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και στην περίπτωση αυτή, αν μιλάμε για τα κράτη-μέλη αυτά θα πρέπει να έχουν την ερμοδιότητα να ε, μπορούν να υλοποιήσουν ένα τέτοιο σύστημα. Μάλιστα, για να κλείσουμε αυτή, αυτή τη δεύτερη, το δεύτερο γύρο, η κυρία Αλφάνο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μάλιστα, καλωσορίζω εδώ όλου του συναδέλφου που εκπροσωπούν ε, εδώ το Εθνικό Κοινοβούλιο. Εγώ είμαι εισηγήτρια για την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οργανωμένο έγκλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για μια έκθεση που εγώ και η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ το έχουμε, την έχουμε υποστηρίξει την έκθεση αυτή και έχει γίνει ένα έργο που συμμετείχαν όλες οι πολιτικές ομάδες ε, και αυτό δεν φάνε από που την ομόφωνη έγκριση στην Επιτροπή Λίμπε στις 29 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για μια έκθεση που αναφέρει ε, τη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουν όλοι οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί ε, και την οργανισμοί. Εκεί περιλαμβάνεται ένας λεπτομερής κατάλογος αιτήσεων και αυτό εξηγείται από το γεγονό ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θέλει να παραμείνει ως ε, παθητικός επέκτης, αλλά θέλει να ασκήσει όλα τα δικαιώματα που του δίνουν οι συνθήκες για το έλεγχο του οργανωμένου εγκλήματος. Επίσης, υπάρχει βούληση να δημιουργηθεί μια επιτροπή κοινοβουλευτική για τη μαφία και για το οργανωμένο έγκλημα προσωρινή επιτροπή, η οποία θα είναι απαραίτητη για να προσδιορίσει τα νομοθετικά και όχι μόνο μέτρα που πρέπει να ληφθούν και για να αναλάβει μια ισχυρή συντονιστική δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εμεί θεωρούμε ότι μέχρι να δημιουργηθεί αυτή η κοινοβουλευτική επιτροπή είναι μακρύ ο δρόμο, ε, αλλά ε, ήδη συνειδητοποιούν όλε οι πολιτικέ ομάδε ότι χρειάζεται μεγάλη αποφασιστικότητα για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο. Εγώ θα ήθελα να αναφέρω ορισμένα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην εκθεσή μα. Αποτελεσματικοί κανόνε για την κατάσχεση ε, των ουσιών που προέρχονται από εγκληματικέ δραστηριότητε. Επίση, η δημιουργία δικτύων κατά τη μαφία στα 27 κράτη-μέλη. Μεγαλύτερο συντονισμό μεταξύ Europol, Eurojust, Olaf και των υπόλοιπων εθνικών αρχών. Βελτίωση τη δικαστική συνεργασία και αναγνώριση πλήρης των δικοστικών αποφάσεων, κανόνες για τη διαφάνεια και την πρόληψη έτσι ώστε ε, δημόσια κονδύλια να μην καταλήγουν στο δίκτυο του οργανωμένου εγκλήματος, κανόνες κατά της ανακύκλωσης ε, του χρήματος, επίσης να αποφύγουμε ε, οι εγκληματίες όσοι έχουν καταδικαστεί ε, για οργανωμένο έγκλημα να μπορούν να θέτουν ψηφιότητα σε ευρωπαϊκές εκλογές, σε ευρωεκλογές. Το ΙΟΚΤΑ, το τελευταίο έγγραφο ανάλυσης για το οργανωμένο έγκλημα, απειλή του οργανωμένο έγκληματος που συντάσσει η Ευρωπόλ. μας δείχνει ότι και το 2011 βλέπουμε μια πολύ ανησυχητική εικόνα και εγώ μπορώ να σας πω ότι ε, υπάρχουν ε, συστηματικές, ε, συγγνώμη υπάρχουν κάποιες περιοχές όπως τα Βαλκάνια, η, η Βαλτική, οι χώρες της Βαλτικής, στην Ιβυρική, στην Νότια Ιταλία βλέπουμε εκεί να δραστηριοποιούνται μαφίες όσα λέγονται στην έκθεσή μας ίσως θεωρούνται δεδομένα, όμως πρέπει να έχουμε κατά νου το εξή, ε, ότι και στα 27 κρατημέλη ε, βλέπουμε πλέον να ριζώνουν εγκληματικέ ε, ομάδε και βλέπουμε ότι υπάρχουν σε διάφορου τομεί στην οικονομία, στη δημόσια δίκηση κτλ όμως ε, κάποια στοιχεία που υπάρχουν στην ΟΚΤΕ δυστυχώς ε, δεν μας οδηγούν σε συγκεκριμένη πολιτική γραμμή για την καταπολέμηση. Σίγουρα ε, έχουμε και κάποια στοιχεία δυτικά όπως σημεία φετηρίας, όπως την ανακοίνωση της Κομισιόν, το Project Harmony και το Project 2012-2013. Αποτελούν αυτά κάποια μικρά βήματα που προωθεί κυρίως το Συμβούλιο και που μας δείχνουν ότι δυστυχώς υπάρχει ελλειπή συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκών εγώ θέλω να υπογραμμίσω ότι εκτιμώ τη δουλειά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κυρίως της Επιτρόπου Μάλστρομ ε, ε, τις προσπάθειες της Europol και της Eurojust ε, να βελτιώσουν τις μεθόδους τις ερευνητικές τους αλλά να σας πω πώς μπορούμε εμείς να παραπονιόμαστε εδώ για την Europol και την Eurojust αν εμείς που εκπροσωπούμε τους πολίτες δεν κάνουμε όσα μπορούμε να πράξουμε δεν βάζουμε τη δυνατά μας δηλαδή πρέπει να δούμε ποιος είναι και ο ρόλος της πολιτικής εγώ νομίζω ότι η απάντηση σε όλα αυτά βρίσκεται στη συνθήκη κυρίως στο άρθρο 10 της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπενθυμίζει ότι η λειτουργία της Ένωσης βασίζεται στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Το άρθρο 12 μιλά για την ενεργή συνεισφορά των Εθνικών Κοινοβουλίων και εγώ πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει από κοινού με τα Εθνικά Κοινοβούλια να αναπτύξει τον ηγετικό του ε, πολιτικό ρόλο και δεν θα πρέπει αυτό ε, να θεωρείται ε, ως παρέκκληση εμείς. Ε, είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να λειτουργήσουμε αποφασιστικά έναντι του οργανωμένου εγκλήματος και η έκθεσή μου αλλά και η έκθεση της συναδέλφου Σοφή Ίντελ ελπίζω να μην παραμείνουν στη θεωρία. Από την ανάλυση θέλουμε να περάσουμε στην πράξη και ελπίζω ότι και ο καθένας να μεταφέρει το μήνυμα μιας κοινή δράση πρέπει να αναλυφθεί από τα Εθνικά Κοινοβούλια και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Με την συνεργασία της Επιτρόπου και επειδή πρέπει να φύγει για να προλάβει το αεροπλάνο της θα δώσω τον ε, λόγο ακόμη στον ε, τελευταίο μιλητή Χάνες Βατζέκα από το Αυστριακό Κοινοβούλιο. Σας παρακαλώ να μας βοηθήσετε με το χρόνο για να μην χάσει το αεροπλάνο της η κυρία Μάλστρομ. Πρέπει 4,5 ώρες ε, να έχει φύγει ο κύριος Βαζέκας. Ευχαριστώ στις ομιλίες από το Προεδρείο τονίστηκε ιδίως ε, η διατήρηση ε, των δικαιο... θεμελιωδών δικαιωμάτων και η προστασία των δεδομένων. Πρέπει να απαντήσουμε στην τρομοκρατία και στην οργανωμένη εγκληματικότητα και γι' αυτό ε, όλο και περισσότερο επεμβαίνουμε στα προσωπικά δεδομένα, στα PNR, στα στοιχεία τα ταξιδιωτικά τα τηλεφωνικά. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω ποια θα είναι η στρατηγική της Ευρώπης τα επόμενα χρόνια εάν ε, ε, η προστασία των δεδομένων υπό το πρίσμα της ε, οργανωμένης εγκληματικότητα πρέπει να διατηρηθεί. Ευχαριστώ που είσαστε σύντομος και δίνω το λόγο στην κυρία Μάλστρομ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ διότι καταρχήν θα ήθελα να πω στον κύριο Μπορσελίνο ότι στο μέλλον θα πρέπει να εστιάσουμε ε, τις εκθέσεις και όταν θα κάνουμε ε, την έκθεσή μας ε, φέτος δεν είχαμε συντονιστεί αλλά όντως του χρόνου θα πρέπει να γίνει μία συνδεδιασμένη συζήτηση για την αξιολόγηση και το ISS. Συμφωνώ Γι' αυτό που είπατε. Η έκθεση είναι εξαιρετική και περιλαμβάνει πάρα πολλά στοιχεία χρήσιμα και πέραν αυτού πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα για να βελτιώσουμε και να συνδυάσουμε την εσωτερική ασφάλεια, να τη συνδυάσουμε με την εξωτερική ε, ασφάλεια και ε, με την κυρία Άστον θα προσπαθήσουμε να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μας με την υπηρεσία εξωτερικής δράσης για να επιλύσουμε ορισμένα προβλήματα όπως το οργανωμένο ε, έγκλημα και την τρομοκρατία συνθήκη όντως προβλέπει ότι πρέπει να υπάρχουν και στρατιωτικά μέτρα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση κρίσεως. Οπότε πρέπει να δούμε πώς θα διαχειριστούμε τις κρίσεις. Αυτό είναι ένα θέμα που δεν έχουμε επεξεργαστεί επαρκώς. Όσον αφορά τον εκπρόσωπο του Γερμανικού Κοινοβουλίου, το PNR τώρα ε, συζητείται με μεταξύ των δύο νομοθετικών θεσμικών οργάνων και θα δούμε πώς θα καταλήξουμε. Βέβαια προσπαθούμε να ενημερώσουμε τους πολίτες και να υπάρχουν μέτρα επανόρθωσης. Θα δούμε πού θα καταλήξουμε τελικά σχετικά με το θέμα αυτό. Όσον αφορά την ε, διαρθρωμένη συνεργασία και ε, ε, το ερώτημα που θέσατε, υπάρχει συνεργασία στα σύνορα Ελλάδος και Τουρκίας και συνεργαζόμαστε με την Τουρκία χωρίς όμως να έχουμε μία δομημένη συνεργασία εσωτερικής ε, ασφαλείας με αυτή τη χώρα. Ε, επίσης ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει αργότερα στο χρόνο μία πρόταση για την δυνατότητα κατασχέσεως των περιουσιακών στοιχείων των εγκληματιών όπως ζήτησε η κυρία Αλφάνο και τέλος σχετικά με τον εκπρόσωπο του Αυστριακού Κοινοβουλίου όντως έχετε δίκιο είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να κοιτάξουμε την αναλογικότητα, την επικουρικότητα είμαστε δεσμευμένοι από τις συνθήκες ε, για να ε, ε, οριοθετήσουμε τα θέματα. Χρειάζεται βέβαια προστασία των προσωπικών στοιχείων και θα διατυπωθεί μία πρόταση για όλους αυτούς οι οποίοι είναι ήδη καταγεγραμμένοι αλλά ήδη μέχρι στιγμής υπήρχαν ορισμένα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιούσαμε παρόλο που πρόκειται για ένα πολύ αμφιλεγόμενο και δύσκολο θέμα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για τη δυνατότητα που μου δώσατε να ανταλλάξουμε τις απόψεις. Πάντοτε χαίρομαι και να συζητώ με τους ευρωβουλευτές αλλά και με τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων για τόσα σημαντικά θέματα. Είναι πολύ χρήσιμο. Σας ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να φύγετε αυτή τη στιγμή για να προλάβετε το αεροπλάνο σας. Σας ευχαριστούμε για τα ε, σχόλιά και δίνουμε το λόγο ή στον ε, ε, Υπουργό κύριο Ραπάτσκι για να σχολιάσει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ στο έργο της μόνιμης ε, Επιτροπής για την Εσωτερική Ασφάλεια στην Κόζη. Γιατί ουσιαστικά θα πρέπει να βρει ποια, ποια είναι τα καθήκοντα που πρέπει να επιτελέσει ε, και αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν επικαλύψεις με τις υφιστάμενες δομές. Ε, πρέπει να επικεντρωθεί στους στρατηγικούς τομείς που να επιτρέψουν ε, την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, την τρομοκρατία, τα προβλήματα που συνδέονται με τη ρήτρα ηλεγγύης και την προστασία των εξωτερικών συνόρων. Επίσης, να διαρθρώσει και την εσωτερική με την εξωτερική ασφάλεια. Όλες αυτές οι προτεραιότητες καθορίζονται στη στρατηγική εσωτερική ασφάλειας ε, και όλα αυτά συζητούνται στην Επιτροπή Κόζη. Η Επιτροπή Κόζη έχει αναλάβει μια μεθοδολογία και έχει οθετήσει μια, μια πολύ συγκεκριμένη μέθοδο εργασίας. Επικεντρώνεται στο οργανωμένο έγκλημα εμείς ε, μελετούμε τις εκθέσεις ε, της Ευρωπόλ και αναλύουμε τις κύριες απειλές που ανακύπτουν ε, από το οργανωμένο έγκλημα. Στη συνέχεια καταρτίζουμε στρατηγικούς στόχους που θέλουμε να πετύχουμε μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα δράσεων. Και με στρατηγικό τρόπο τι κάνουμε. Προετοιμάζουμε ένα πρόγραμμα δράσεων που συνάδουν με όσα γίνονται στις υπόλοιπες υπηρεσίες και οργανισμούς της Ένωσης και με όσα γίνονται στις διάφορες εθνικές υπηρεσίες. Αυτό που κάνουμε είναι να επικεντρωνόμαστε στους κύριους τομείς ε, καταπολέμησης ε, των κυρίων εγκλημάτων. Φυσικά δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με τα πάντα. Έτσι λοιπόν προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τους τομείς όπου πιστεύουμε ότι χρειάζεται ανάληψη δράσης. Και στον ε, κύκλο προγραμματισμού του χρονοδιαγράμματος αυτό που κάνουμε είναι να αναλύουμε τις συνέπειες ε, και να βλέπουμε ποια συμπεράσματα μπορούμε να ξαγάγουμε για να επιλύουμε τα διάφορα προβλήματα που προκύπτουν από την εγκληματικότητα, κυρίως Βλέπουμε πώς μπορούμε επίσης να προσεγγίσουμε την εσωτερική πολιτική με την εξωτερική πολιτική και με τις υπόλοιπες πολιτικές όπως είναι η πολιτική γειτονία. Επίσης προετοιμάζουμε ένα χάρτη πορείας που θα συζητηθεί στο ιστορικό της Κόζη και μαζί με την Κομισιόν θέλουμε να προετοιμάσουμε μία μέθοδο δράσης και ένα πρόγραμμα λύσεων. Αυτές είναι ήδη συγκεκριμένες δράσεις που από στρατηγική σκοπιά οικοδομούν όλο αυτό το σύστημα εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Παρακαλώ, θέλετε να πάρετε το λόγο. Κύριε Μπορσελίνο. Ναι. Αυτό που προέκυψε από τις διάφορες ε, παρεμβάσεις νομίζω ότι μπορεί να συνοψιστεί με δύο λόγια. Είναι πολύπλοκες οι κυρίες έννοιες, θεμελιώδεις έννοιες, αλλά μπορούμε να τις προσδιορίσουμε με δύο λόγια. Η έννοια της ασφάλειας δεν ε, μπορεί να ε, διαφοροποιηθεί από την έννοια του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων το να θέτουμε από κοινού αυτά τα δύο είναι κάτι ιδιαίτερα πολύπλοκο, αλλά είναι κάτι απολύτως απαραίτητο. Ένα άλλο στοιχείο που ανακύπτει είναι το θέμα της αναγκαιότητας να εργαστούμε από κοινού. Δηλαδή να έχουμε, συνεργασία όχι μόνο με τα εθνικά κοινοβούλια, αλλά να συνεργαζόμαστε και με την Κομισιόν και με τους οργανισμούς και με το Συμβούλιο είναι δυνατόν. Γιατί ένα τέτοιο τόσο πολύπλοκο και σημαντικό θέμα χρήζει συνεργασίας που να έχει ως ε, στόχο την ε, ασφάλεια, την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών. Αναφέρθηκε και το θέμα της ασφάλειας ε, και των δικαιωμάτων των πολιτών τρίτων χωρών. Εμείς ε, ακούσαμε ότι αναφέρθηκαν κάποιοι στην ε, αναγκαιότητα να εκπονηθούν και κανόνες, να εκπονηθεί και νομοθεσία. Αυτό ουσιαστικά προκύπτει από ε, την αξία της αλληλεγγύης, που είναι μια θεμελιώδης αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει ασφάλεια αν δεν υπάρχει αλληλεγγύη και δεν ε, σκοπεύω εγώ να απομακρυνθώ από την έννοια αυτή στο έργο μου. Μάλιστα, ευχαριστούμε την κυρία Μπορσελίνο, ο καθηγητής Κατάλντι. Μάλιστα, πολύ γρήγορα. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με την προηγούμενη παρέμβαση οι οργανισμοί από τεχνική σκοπιά και υπηρεσιακή σκοπιά ε, συνεισφέρουν τα μάλλα. Εγώ γνωρίζω πολύ καλά πώς λειτουργεί η Frontex, γιατί έχω συνεργαστεί με τη Frontex, όμως είναι προφανές ότι όλα όσα γίνονται θα πρέπει πάντοτε να γίνονται με έναν ισορροπημένο τρόπο. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ θεμελιωδών δικαιωμάτων και αποτελεσματικότητας. Και στην Ευρώπη είδαμε ότι υπήρχε καλή ισορροπία μεταξύ σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη ασφάλεια ε, που χρειαζόμαστε μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Ανελήφθησαν κάποιε πρωτοβουλίε, ε, οι οποίε ορισμένε φορέ ε, δέχτηκαν και κριτική είτε από τα εθνικά κοινοβούλια είτε από τα δικαστήρια. Αυτό έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ιταλία, στη Γαλλία. Και αυτή είναι η ορθή λειτουργία μια δημοκρατία. Τώρα η Ευρώπη, είναι προφανές ότι η Ευρώπη έχει μεγάλες ευθύνες. Εμείς ε, έχουμε ένα ελάχιστο ε, πρότυπο να σεβόμαστε τα δρόμινα δικαιώματα. Αυτό δεν είναι διαπραγματεύσιμο. Ε, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να το καταλήψουμε και αυτό είναι σημαντικό και συχνά στο πλαίσιο της διεθνούς κοινότητας ε, πολλές φορές ε, βλέπουμε ότι όταν γίνεται μια προσπάθεια καταπολέμησης της πειρατείας στη Σομαλία ε, τότε δίνει η διεθνής κοινότητα στην Κένια την δικαιοδοσία να δικάσει τους πειρατές έχω κάποια αμφιβολία εγώ. Δηλαδή έχουμε εκεί συλλογική ευθύνη γιατί δεν ξέρουμε σε ποιον ουσιαστικά πρέπει να γίνει αυτή η λογοδοσία. Και έτσι λοιπόν ξέρουμε ότι το σύστημα της Λισαβόνας ότι αφορά ε, το, αρμοδιότητα ε, για τον έλεγχο των οργανισμών αυτών ακόμη δεν έχει υλοποιηθεί γιατί μας λείπει από την πλευρά της Κομισιόν μια πρόταση για το πώς μπορούμε να δράσουμε. Και ε, ίσως τελικά μπορούμε να καταλήξουμε στο να μην ξέρουμε ποιος είναι υπεύθυνο και με ποιο τρόπο. Και αν ε, χρειαστεί, αν βρούμε κάποιο υπεύθυνο, πώς θα τον οδηγήσουμε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, σύμφωνα με ορισμένα άρθρα των συνθήκων, γιατί ακόμη δεν υπάρχει αυτός ο σύνδεσμος που σας είπα προηγουμένως. Και φυσικά όταν μιλάμε για μετανάστευση, η μετανάστευση είναι ένα δεδομένο, δεν μπορούμε να το εξαλείψουμε, πάντοτε υπήρχε στην ιστορία της ανθρωπότητας. Έτσι λοιπόν ε, μιλάμε απλώ για τη διαχείριση ενός φαινομένου. Δεν ε, είναι ένα πρόβλημα, είναι ένα δεδομένο το οποίο πρέπει να έχουμε κατά νου δεν υπάρχει άλλη οδό στι δημοκρατίες στα ευρωπαϊκά κράτη. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε εδώ κάποιες εκτόσει απλώς επειδή έχουμε ένα οικονομικό πρόβλημα γιατί η ισχύ ενός δημοκρατικού συστήματος ε, αποδεικνύεται τη στιγμή της δυσκολίας. Ωραία. Χωρί περαιτέρω καθυστέρηση ευχαριστούμε τα μέλη του πρώτου γύρου και θα αρχίσουμε αμέσως το δεύτερο τμήμα που λέγεται πρώτο στο πρόγραμμα για την πρόληψη και καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και το ρόλο επ' αυτού της Ευρωάστρα. Πρώτος ομιλητής, ο κύριος Ρομπ Βουέινράιτ, διευθυντής της Ευρωάστρα και μετά θα μιλήσουν και άλλοι. Ευχαριστούμε λοιπόν τους πρώτους και καλωσορίζουμε τον κύριο Rob Wainwright. Σαν πως θα το ακολουθήσει. Λέει ότι το Just, just a second. Yes. Ο κύριος Δίας Δεμέρα θα μιλήσει μετά τον κύριο Ρομπ Wainwright. Γιατί έχει γίνει μια αντικατάσταση για ιατρικούς λόγους. θα αντικατασταθεί από τη συνάδελφο Τερέσα Χιμένης Πλησερέιδου που θα μιλήσει εξ ονόματος της Επιτροπής Ελευθεριών, Δημοσίων Ελευθεριών. Για τους εφαρμοστικούς κανόνες των αναλύσεων που κάνει η Ευρωάστ και μετά θα μιλήσει ο καθηγητής Γιώργ Μόναρ διευθυντής σπουδών στο Κολέγιο της Ευρώπης Πρώτα πρώτα όμως όπως προείπα θα μιλήσει ο διευθυντής της Europol ο κύριος Rob Wainwright. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτέ του Ευρωπαϊκού και των Εθνικών Κοινοβουλίων, σας κατευχαριστώ για την πρόσκληση της Ευρωπόλ σε αυτή τη συνάντηση για να συζητήσουμε την δημοκρατική λογοδοσία γιατί νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό στοιχείο στη συζήτησή μας. Θα ήθελα σήμερα να σας παρουσιάσω τι έχουμε παρατηρήσει στην Ευρωπόλ με τα Εθνικά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να μοιραστούμε ορισμένες σκέψεις για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε στην πράξη να εφαρμόσουμε δημοκρατική λογοδοσία. Πρώτα πρώτα θα γνωρίζετε ότι η Ευρωπόλ είναι το κύριο όργανο της Ένωσης για την επιβολή της ένωμης τάξης. Συντονίζουμε, προσπαθούμε να έχουμε μια συντονισμένη ανταπόκριση στη σοβα... στα σοβαρά εγκλήματα και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στην Ευρώπη. Διευκολύνουμε τις ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ τελωνιακών και άλλων αρχών. Η αυτής μεγαλειώτης η βασίλισσα της Ολλανδίας την 1η Ιουλίου εφέτος εγγενίασε τα, τη νέα μας έδρα και η οποία στεγάζει 700 εμπειρογνώμονες και αναλυτές καθώς και συντονίζει 14.000 περίπου έρευνες κάθε χρόνο. Οι υπηρεσίες και τα όργανα ολόκληρης της Ένωσης δεν έχουν διοκτικές δικαιοδοσίες αλλά μπορούν να βοηθήσουν στη διαλεύκανση πολλών ερευνών και εγκλημάτων. Επίσης φυσικά συνεργαζόμαστε και με άλλες ευρωπαϊκές υπηρεσίες όπως το Ευρω... την Eurojust και το Frontex καθώς και διεθνώς συνεργαζόμαστε με την Interpol και με υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχουμε επαναλαμβάνω διοκτικές δικαιοδοσίες αλλά νομίζουμε ότι οι δυνατότητες μας πολέμηση στο εγκληματικότητα έχουν διευκολύνει πολλές έρευνες και οδήγησαν στην σύλληψη πολλών επικινδύνων εγκληματιών τελευταία καθώς και εκατοντά, βοήθησαν εκατοντάδες θυμάτων δουλεμπορίου συμπεριλαμβανομένων και παιδιών. Όπως θα γνωρίζετε μετά από αυτά που έγινε στην Ορβηγία στις 22 Ιουλίου η Ευρωπόλα άρχισε να λειτουργεί το πρώτο δίκτυο ανταπόκρισης για να διευκολύνει τις χώρες μέλη να στηρίξουν όσους είχαν αναλάβει την έρευνα στην Νορβηγία και να κάνει μια αξιολόγηση της απειλής που αντιπροσωπεύουν οι εξτρεμιστικές ενέργειες. Άλλο πρόσφατο παράδειγμα της πρόσθετης αξίας της δουλειάς μας είναι η περσινή Operation Rescue, η μεγαλύτερη περίπτωση εκμετάλλευσης παιδιών. Οι αναλυτικές μας δυνατότητες οδήγησαν στην ταύτιση 705 υπόπτων, από τους οποίους σχεδόν 200 συνελήφθησαν. και ταυτίστηκαν επίσης 230 παιδιά ως θύματα. Τώρα, ως προς τις εσωτερικές δομές ασφαλείας της Ένωσης, αυτό έχει αποσαφινιστεί χάρη στις προτεραιότητες και τη στρατηγική που καθορίστηκαν από την Ευρώπη με την συντονισμένη διαδικασία αξιολόγησης που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις πληροφορίες που συλλέγουμε από τις χώρες μέλη. και με βάση αυτές τις πληροφορίες καταστρώνονται στρατηγικές για να βρε... καθορίσουμε προτεραιότητες. Από τη δεκαετία του 90 περάσαμε σε μια πλήρη ευρωπαϊκή υπηρεσία για πρώτη φορά. Έχει συζητηθεί πολύ το θέμα των ευθυνών που πρέπει να αποδίδονται στην Ευρωπόλ και η συνθήκη της Λισαβόνας φυσικά βάζει το Ευρωπαϊκό και τα Εθνικά Κοινοβούλια στην καρδιά της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και σε αυτό το θέμα πράγμα που συνδυάζεται με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που ενέκρινε η Ευρώπη πρόσφατα. Αυτό οδήγησε σε αύξηση των δικαιοδοσιών της Ευρωπόλ Είμαστε υπεύθυνοι στα μάτια του Διοικητικού μας Συμβουλίου αλλά επίσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που από κοινού για πρώτη φορά είναι αρχές συνυπεύθυνες για τον προϋπολογισμό μας. Συμβουλευόμαστε πάρα πολλά νομοσχέδια τα οποία αναλύουμε. Εγώ ίδιος πηγαίνω συχνά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και έχω επισκεφθεί και πολλά εθνικά ιδιαίτερα από την Βρετανία, Ιταλία, Ισπανία και Γερμανία που επιδεικνύουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη δουλειά μας. Όπως είπα και πριν, το νομικό πλαίσιο της λειτουργίας μας έχει αλλάξει από το 2010 μετά τη θέση ενισχύτηση της συνθήκης της Λισαβόνας έτσι ώστε να είμαστε πιο δημοκρατικά υπόλογοι. Εδώ ο ρόλος του Κοινοβουλίου δεν περιορίζεται μόνο στον προϋπολογισμό αλλά και στην επιτήρηση και εποπτεία της λειτουργίας της Ευρωπόλου. Η Κομισιόν μάλιστα πρότεινε μια νέα νομική βάση, ένα νέο νομικό υπόβαθρο, το άρθρο 88 της Συνθήκης Λισαβόνας για τη λειτουργία της Ευρωπόλου. Νομίζουμε ότι αυτό είναι μεγάλη ευκαιρία να βελτιώσουμε περαιτέρω το δημοκρατικό χαρακτήρα της Ευρωπόλου ώστε η υπηρεσία αυτή να είναι και πιο αποτελεσματική στη δουλειά της. Ανεξάρτητα ανεξάρτητη αξιολόγηση της δουλειά μας αυτή τη στιγμή γίνεται και θα αναφερθεί στα μέλη του Κοινικού μας Συμβουλίου. Από τα συμπεράσματα θα πάρουμε μαθήματα που νομίζω θα είναι πολύ χρήσιμα για το μέλλον μας. Αυτή νομίζω θα είναι η τελευταία μεγάλη αναδιοργάνωσή μας έτσι ώστε να σταθούμε στο ύψος των απαιτήσεων που έχει η Ένωση από μας. Ποιες είναι οι βελτιώσεις. Πρώτον, η Ευρωπόλ θα μπορεί να δίνει μεγαλύτερη χρηματική στήριξη σε ορισμένες έρευνες. Είναι κάτι που έχουμε δικαίωμα να το κάνουμε για να υπάρχει παραγωγικότερη χρήση του χρηματοδοτικού μηχανισμού της Ένωσης. Επίσης, να αναπτυχθούν οι δυνατότητες μας περιφερειακής στήριξης των προσπαθειών των χωρών μελών για την καταπολέμηση των κυρίων επικέντρων του οργανωμένου εγκλήματος ολόκληρη την Ευρώπη. Επίσης νομίζω ότι μπορούμε να βασιστούμε στην θετική μας εμπειρία ως κεντρικού οργάνου πρόληψης και καταπολέμησης των... της παραχάραξης των ευρώ. Εκτός από αυτά τα πιο συγκεκριμένα θέματα προβλέπεται ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ Ευρωπόλ και Εθνικού και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίων. Πολλές φορές γίνεται λόγος για εξισορρόπηση μεταξύ υπολογισμότητας συλλογίας και υπολογισμότητας μάλλον και αποτελεσματικότητας. Είναι πράγματι ένα πρόβλημα αυτό. Πρόσφατα υπόθηκε στον τύπο ότι Μπορεί η Ευρωπόλ να έχει αρκετά περιορισμένη αποτελεσματικότητα, αλλά θα βελτιωθεί αυτό στο μέλλον. Η τελευταία αναφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την επιτήρηση της λειτουργίας της Ευρωπόλ δήλωνε ότι είναι ίσως η πιο ελεγχόμενη αστυνομική αρχή στην Ένωση. Και ακούστηκε έπαινος των δραστηριοτήτων μας ως προτύπου για τις αστυνομικές δραστηριότητες στην Ένωση. Βέβαια και εδώ υπάρχει χώρος βελτίωσης και φαντάζομαι θα τα πείτε και εσείς στη συζήτηση όπως κάναμε και με την Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών τους τελευταίους μήνες. Ορισμένες πρακτικές ιδέες όμως. Πρώτον, η συνεργασία με τους ευρωβουλευτές και τους εθνικούς βουλευτές θα μπορούσε και αυτή να ενδυναμωθεί χορηγώντας περισσότερη πληροφόρηση για τις δραστηριότητες μας τον Απρίλιο οι ευρωβουλευτές πήραν μία έκθεσή μας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και τακτικά τους στέλνουμε απολογισμούς και αξιολογήσεις για την καταπολέμηση του οργανωμένου κλίματος. Επίσης γίνεται μία γενική έκθεση των δραστηριοτήτων της Ευρωπόλ πιστεύω ότι τέτοιου είδους εκθέσεις και αναφορές θα έπρεπε να υποβάλλονται και στην ΚΟΖΑΚ. Εν τω μεταξύ, τακτικές συναντήσεις διοργανώνονται με τους αξιωματούχους της Ευρωπόλ και τους Ευρωβουλευτά για περισσότερη αμοιβαία κατανόηση. Νομίζω ότι οι συναντήσεις που έγιναν και με εθνικούς βουλευτές και πολλά μέλη της Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών πάντοτε υπήρξαν επικοδομητικές ως ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών. Και χαίρομαι ιδιαίτερα, θα χαιρόμουν ιδιαίτερα να ερχόμουν ακόμη συχνότερα στο Κοινοβούλιο από ό,τι γίνεται μέχρι τώρα. Επίσης πιστεύω ότι θα μπορούσε να αυξηθεί κατανόηση της αξίας της δουλειάς της Ευρωπόλ μέσω της δημιουργίας μιας υποεπιτροπής της Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών που να ασχολείται ειδικά με αυτό το θέμα. Αυτό το πρότεινε τελευταία σε ένα ψήφισμά του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για να καταλήξω η επιβολή του νόμου και της τάξης είναι από τα θεμελιώδη δικαιώματα και είναι εγγύηση της εφαρμογής τους. Η Ευρωπόλ χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαίο Φορολογούμενο και την Ευρωπαία Φορολογούμενη και επομένως είναι υποχρεωμένη να έχει διαφανή λειτουργία και οτιδήποτε μπορεί να βελτιώσει τη διαφάνεια αυτή θα το δεχτούμε. Δεχόμαστε ιδιαίτερα όλες τις συμβουλές των βουλευτών και ευρωβουλευτών για περισσότερο αποτελεσματική εργασία και πιστεύω ότι ο νέος μας κανονισμός βελτιώνει τα πράγματα και ως προς τη διάσταση αυτή καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να, να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη για να καταπολεμήσουν την τρομοκρατία. Άρα τελικά η λογοδοσία είναι τρόπος βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και για την ταύτιση και δίωξη των εγκληματιών ώστε η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει μια ασφαλέστερος χώρος. Ευχαριστώ ιδιαίτερα κύριε Πρόεδρε τους Ευρωβουλευτάς και τους Βουλευτάς για τη συνεργασία μας. Ευχαριστώ. Τώρα θα ακούσουμε την κυρία Χιμάνη Πεσερίλ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καλησπέρα σας. Είναι τιμή μου να περιβρίσκομαι εδώ ενώπιόν σα. Όπως βλέπετε, εγώ δεν είμαι ο κύριος Αγκουστίν Δίας Δαμέρα, γιατί αναγκάστηκε να απουσιάσει, γιατί είχε ένα πρόβλημα στην Ισπανία. Αλλά συνεργάζομαι μαζί του στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και όπως και αυτός έχω και εγώ φιλοδεξία να καταπολεμήσουμε όλα τα εγκλήματα και την τρομοκρατία. Ασχολούμαι γενικά με θέματα υπεράσπισης των θυμάτων. Τώρα συντάσσω μια έκθεση για την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας. Πρόκειται για το νέο νομοθέτημα για τα θύματα που προετοιμάζουμε. Πάντω, βρίσκομαι εδώ για να μιλήσω για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο των δραστηριοτήτων τη Europol, τη συνθήκη τη Λισαβόνα και τη μελλοντική πρόταση κανονισμού. Στο στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 88 της Συνθήκης της Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλώνεται ότι το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα καθορίσουν μέσω κανονισμών που θα έχουν θετηθεί σύμφωνα με την τακτική νομοθετική διαδικασία συναπόφαση, την δομή, τη λειτουργία, το πεδίο δράσης και τις αρμοδιότητες της Ευρωπόλ. Αυτή η διαδιάταξη προβλέπει ότι στο μελλοντικό κανονισμό θα θεσπίζονται διαδικασίες ελέγχου της δραστηριότητας της Ευρωπόλ από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έλεγχος στον οποίο θα πρέπει να συμμετάσχουν και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Το σημερινό ρυθμιστικό πλαίσιο της Europol δεν προβλέπει ένα πραγματικό μηχανισμό δημοκρατικού ελέγχου των δραστηριοτήτων της. Τα μέτρα που αναφέρονται στην απόφαση της Europol περιορίζονται στον δημοσιονομικό έλεγχο. Πρόκειται για το άρθρο 42 και το άρθρο 43 της απόφασης του Συμβουλίου αποκλείοντας ε, κάθε δυνατότητα να ελαιοποιηθεί ένας πραγματικό κοινοβουλευτικό έλεγχος ε, των δραστηριοτήτων ε, του οργανισμού. Η απόφαση του Συμβουλίου φαίνεται να θέσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, φαίνεται να στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μία θέση απλώ παρατηρητή και όπω ξέρετε συμβουλευτικές λειτουργίες δεν έχουν κανένα πραγματικό αποτέλεσμα. Η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, θέτει διάφορα ζητήματα σε ένα έγγραφο που σίγουρα θα οδηγήσουν ε, σε ε, κάποια επίμαχα ζητήματα. Η εν λόγω έκθεση αναφέρει τις τεχνικές και επιχειρησιακές δυσκολίες που σχετίζονται με έναν υποθετικό κοινοβουλευτικό έλεγχο των δραστηριοτήτων της Europol και των λοιπών υπηρεσιών του χώρου ελευθερίας δικαιοσύνης και ασφάλεια Μεταξύ άλλων ε, ζητημάτων ε, αναφέρονται και λόγοι σχετικά με το απόρριτο την ε, δυνατότητα παρέμβαση σε αρμοδιότητε εθνικού χαρακτήρα, οι πιθανέ αρνητικέ συνέπειε για την αποτελεσματικότητα τη λειτουργία των οργανισμών και που θα μπορέσουν να επέλθουν αν μια επιτροπή κοινοβουλευτική προβεί σε έλεγχο και ουσιαστικά για την ε, Ευρωπόλη και την Ριοστάση θα αναφέρεται αυτή την αρμοδίση για την προστασία των ε, δεδομένων. Έτσι λοιπόν, τώρα δίνεται μια πραγματική ευκαιρία έτσι ώστε αυτό το κοινοβούλιο να μπορέσει να συμμετέχει ε, στην εποπτεία των δραστηριοτήτων της Europol η συζήτηση που υλοποιούμε τώρα θα πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε για να συγκρουμήσουμε ποια μέτρα ελέγχου μπορούν να υλοποιηθούν για τις δραστηριότητες ε, της ε, Europol. Σε ό,τι αφορά πέρα από ό,τι προβλέπετε ε, για την προστασία των δεδομένων. Εγώ θα έλεγα ότι για το Κοινοβούλιο αυτό είναι θεμελιώδης η ορθή λειτουργία της Europol και όλων των οργανισμών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό καθίσταται σαφέ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει έναν εποπτικό ρόλο όλων αυτών των δραστηριοτήτων και επομένω είναι θεμελιώδη αυτό ο μελλοντικό κανονισμό, είναι απαραίτητο να υπάρχει εμπιστοσύνη. Εγώ πιστεύω, όπω ε, είπε και ο Γουέιν Ράιτ, ε, είναι πολύ σημαντική αυτή η εμπιστοσύνη γιατί αποτελεί τη βάση μια καλή συνεργασία και όπω είπε και ο διευθυντή, αυτό μπορεί να βελτιωθεί με καλύτερη ενημέρωση από την πλευρά του οργανισμού. Εγώ νομίζω ότι σε θέματα ασφάλειας είναι σημαντική η ανταλλαγή πληροφοριών γιατί αυτή είναι η κινητήρια δύναμη και ε, τα εκεί πρέπει να κατευθυνθούμε. Αν ε, εμείς δεν κατορθώσουμε να πετύχουμε το στόχο αυτό, τελικά αυτοί που θα κερδίσουν θα είναι οι τρομοκράτες και οι εγκληματίες. Και φυσικά εμείς δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Μπεσερίλ. Και τώρα για να ολοκληρώσουμε τις παρεμβάσεις ε, του πάνελ και να ξεκινήσει η συζήτηση θα ακούσουμε τον καθηγητή Γιώργ Μόναρ, ε, ο οποίος είναι διευθυντής μελετών στο Κολέγιο της Ευρώπης. Παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, και αξιότιμοι ευρωβουλευτές είναι μεγάλη τιμή για μένα ε, να ε, συμμετέχω σε αυτή τη συνεδρίαση σήμερα το απόγευμα με στόχο να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία και θα εξετάσω το κάθε ένα από αυτά τα θέματα διότι από πλευράς αξιολογήσεως δεν υπάρχει ε, ε, καμία αμφιβολία ότι ε, υπάρχει μία αξιολόγηση της, της κατανοήσεως των διασυνοριακών απειλών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε, έχει περάσει πολύ καιρός από τότε όπου ο κύριος Στόμπεκ μου είχε πει ότι μαθαίνει τις πληροφορίες από τις εφημερίδες διότι τα κράτη-μέλη δεν τον ενημέρωναν επαρκώς. Πιστεύω όμως ότι τώρα ότι η Ευρωπόλ κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να ενημερώνει και ενδεχομένως μπορεί να μιλάμε ε, για την τεχνική πλευρά της Europol είναι όμως μια οργάνωση που είναι και πολύ πολιτική γιατί μόνο έτσι μπορεί να καταρτήσει πολιτικές προτεραιότητες και στον ε, νέο κύκλο πολιτικής ε, οι αξιολογήσεις της Ευρωπόλ θα είναι ακόμη πιο σημαντικές για να εντοπίσουν τις προτεραιότητες. Εδώ θα ήθελα να είμαι κάποιος πιο κριτικός διότι αυτό το οποίο δεν έχουμε ακόμη στην αξιολόγηση αυτή των εγκλημάτων είναι το κόστος των εγκλημάτων ε, σε σχέση με το ε, ανθρώπινο ε, κόστος δηλαδή τον αριθμό των θυμάτων βλέπουμε ότι σε κάθε χώρα υπάρχει ένα κόστος για την ε, εμπορία ανθρώπων και υπάρχουν και πολλά οικονομικά, ε, ε, οικονομικές δαπάνες πέραν των άλλων οι δαπάνες οι οποίες καλύπτονται από τους φορολογουμένους. Εάν λοιπόν η Europol μπορούσε να περιλάβει αυτά τα στοιχεία κόστους των διαφόρων μορφών εγκλημάτων θα ήταν πολύ χρήσιμο διότι δεν έχουμε μεν επαρκή στοιχεία επ' αυτού αλλά πρέπει να έχουμε μία σαφή εικόνα για το ποιο είναι το κόστος για την κοινωνία για τους πολίτες μας διότι θα αντιμετωπίσουμε πολύ σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα και χρειαζόμαστε σε εθνικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά ε, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να γνωρίζουμε πώς θα έχουμε τα μέσα να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα και άρα ποιος είναι ο βασικός ποιο, είναι το βασικό κόστος ε, της καταπολέμησης. Πέραν όμως αυτό υπάρχει και το θέμα της προλήψεως διότι η Europol ε, συμβάλλει στην καταστολή του οργανωμένου εγκλήματος αλλά στο άρθρο 5 παράγραφος 4 της αποφάσεως του Europol η οργάνωση αυτή μπορεί ε, να έχει μία πιο ενισχυμένη εντολή στον τομέα της προλήψεως εγκλημάτων ε, έχοντας ε, περισσότερη εμπειρία και υπάρχει στην Ευρώπη ένα μεγάλο ε, υπάρχουν πολλές δυνατότητες να συγκεντρώσει κανείς εμπειρογνώμονες και μπορούμε να δούμε πώς μπορούν να προληφθούν διάφορα εγκλήματα. Ορισμένες χώρες έχουν περισσότερη εμπειρία σε ορισμένους ε, τομείς την οποία θα μπορούσαν να μεταδώσουν και σε άλλες χώρες. Και κατά αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι Υπάρχει εντύπωση εις ε, το κοινό ότι η Ευρωπόλη είναι ιδίως κατασταλτική οργάνωση ενώ θα έπρεπε να τονίσουμε και τον προληπτικό χαρακτήρα της δράσεώς της βέβαια δεν έχει καταναγκαστικές ε, αρμοδιότητες και η καταστολή αναλαμβάνεται από τις εθνικές αστυνομικές αρχές αλλά βρίσκεται η Ευρωπόλ στην πρώτη γραμμή της καταπολέμησης της τρομοκρατίας γιατί καμία οργάνωση ε, δεν είναι πιο κατάλληλη για να αξιολογήσει πώς μπορεί να οργανωθεί ε, ε, διασυνοριακά η επικοινωνία και η συνεργασία των εθνικών αρχών περισσότερο και από την Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο ή ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άρα θα μπορούσε ε, να εντοπίσει η Ευρωπόλ ορισμένους τομείς ελληματικούς, καλύτερα από ότι άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ε, αντιλαμβάνομαι ότι η Ευρωπόλ πάντοτε δεν θεωρείται ότι πάντοτε είναι πολύ αποτελεσματική και επιπλέον ζητάμε να είναι και διπλωματική. Ε, πρέπει λοιπόν να κινηθεί πάρα πολύ προσεκτικά για να αποφύγει ε, τις ευθυξίες των διαφόρων χώρων αλλά ε, γνωρίζει ίσως η νομοθεσία χρειάζεται ακόμη για να καταργηθούν τα προσκόμματα στη διασυνοριακή συνεργασία ε, αυτό δεν μειώνει το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην πρόταση, νομοθετικ... στην ε, πρόταση νομοθετικών ε, προτάσεων αλλά στην... βοηθά στην καθοδήγηση. Επίσης δεν υπάρχει συγκεκριμένη εντολή προς την Europol προς αυτή την κατεύθυνση. Έχει όμως την εμπειρία και μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη των αστυνομικών δυνάμεων σε ορισμένες χώρες. Οπότε πρέπει να αναρωτηθούμε. Εάν βελτιώσουμε τους εμπειρογνώμονες σε ορισμένες χώρες θα χρησιμοποιηθεί η εμπειρία αυτή για το σωστό σκοπό ή υπάρχει ο κίνδυνος ε, η εμπειρία αυτή να χρησιμοποιηθεί για καταστολή που δεν συνάδει με τις δημοκρατικές αρχές μας αλλά ε, εάν κοιτάξουμε σφαιρικά όλα τα κράτη-μέλη και ιδίω τις επαφές της Europol με τρίτες χώρες ε, θεωρώ ότι είναι σε μία μοναδική θέση και γι' αυτό υπάρχουν τα ε, έγγραφα κάθε εξάμεινο του Διευθυντή της Europol για την καταπολέμηση παραδείγματος χάρη της οργανωμένης τρομοκρατίας Εάν λοιπόν μπορεί να χρησιμοποιήσει η Europol τις δυνατότητές της να ξεκινήσει ε, μία συζήτηση επενός θέματος θα μας βοηθούσε πάρα πολύ όλους. Επίσης ε, ε, είδα τους διάφορους δείκτες αποδόσεως και επιδόσεων και με εντυπωσίασαν. Βλέπετε ότι η Europol προσπαθεί να κάνει ό,τι δυνατόν καλύτερο με περιορισμένα μέσα και ο, ε, φέτος ο προπολογισμός σας ήταν πολύ περιορισμένος. Πρέπει λοιπόν να πιέσει για να μπορέσει το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να της διαθέσει περισσότερους φόρους. Δεν μπορεί κανείς να παγώνει έναν προπολογισμό αλλά όλοι μπορούμε να πούμε ότι η Europol δεν θα μπορέσει να αντεπεξέλθει ε, την αύξηση των ε, καθηκόντων που της ανατίθενται χωρίς ε, να ζητήσει κανείς από τα κράτη-μέλη να αναβαθμίσουν την προτεραιότητα των πόρων που τις διαθέτουν. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να βοηθήσει στο σημείο αυτό. Τώρα όσον αφορά τους δείκτες αποδόσεως. Ε, ίσως ξέρετε ότι τα αγγλικά πανεπιστήμια έχουν ε, μία έμονη ιδέα με, αυτές, με αυτούς τους δείχτες και όλοι προσπαθούν να παρουσιάσουν ε, υπό την καλύτερη δυνατή γωνία τις επιδόσεις τους, να φουσκώσουν τα νούμερα ώστε να φαίνονται καλύτερα. Ελπίζω ότι δεν έχετε τέτοιο κίνδυνο, δηλαδή ότι εδώ θα δείτε να φουσκώνουν τα στατιστικά στοιχεία και συγχρόνως αυτό δεν θα αφαιρέσει σημαντικούς πόρους που μπορούν να ασχοληθούν με πιο σημαντικά θέματα. Δηλαδή ε, καλύτερα είναι να ασχοληθεί κανείς με την ουσία και όχι με τους στατιστικούς στόχους. Τέλος, όσον αφορά τη συνεργασία της Europol με το Κοινοβόλιο, είναι πολύ σημαντικό για την νομιμοποίηση του χώρου της ε, ελευθερίας της ε, ε, δημοκρατίας και ασφαλ... δικαιοσύνης και ασφαλείας να ε, ενισχύσουμε την Ευρωπόλ και να την αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά και το Κοινοβούλιο. Διάβασα όμως εις την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Δεκεμβρίου του 2010 κάτι που με ανησύχησε γιατί λέγεται ότι θα κατατιστούν προτεραιότητες για τις ενέργειες του οργανισμού. Εγώ νομίζω ότι ήδη υπάρχουν πολλές προτεραιότητες που έχουν καταρτιστεί από τα κράτη-μέλη και αποστέλλονται στην Ευρωπόλ. Εάν όμως τα εθνικά κοινοβούλια καταρτίζουν τις δικές τους προτεραιότητες και ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άλλες, τότε ε, ενδέχεται να περιπλακεί η κατάσταση διότι η Ευρωπόλ είναι ένα εκτελεστικό όργανο Καλύτερα λοιπόν να κάνετε ε, ερωτήσεις στην Europol, να ερευνήσετε και αν δεν ικανοποιηθείτε να την κατακρίνετε. Αλλά αφήστε να καταρτήσουν μόνοι τους τον κατάλογο προτεραιοτήτων τους γιατί νομίζω ότι αυτό θα είναι πιο αποδοτικό κατά τη δικιά μου άποψη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα λοιπόν μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις, προτάσεις, συστάσεις. Η ε, Εθνική Βουλή ε, βουλευτές ή οι ευρωβουλευτές. Ο κύριος Σανταμαρτίνη από το Ιταλικό Κοινοβούλιο είναι πρώτος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι τιμή μου που παραμβαίνω σε αυτήν την ακρόαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα ήθελα να στραφώ κυρίως στον επικεφαλής ε, της ε, Europol για να κάνω μία ερώτηση. Ποια πολιτική υλοποιεί η Europol ε, για να προσπαθήσει να καλλιεργήσει ένα κοινό πολιτισμό, μια κοινή κουλτούρα σε σχέση με τις έρευνες των αστυνομικών αρχών και κυρίως ε, σε ό,τι αφορά ε, τα διάφορα συστήματα των κρατών μελών, ε, κυρίως σε ό,τι αφορά τη συλλογή των αποδεικτικών στοιχείων. Έχουμε υπόψη ότι πολλές φορές όταν μιλάμε για θέματα που μας αφορούν σε σχέση με την καταπολέμηση τρομοκρατίας του οργανωμένου εγκλήματος, δεν λαμβάνονται υπόψη διαφορετικές λειτουργίες ε, και καθήκοντα έχουν οι δημόσιοι κατήγοροι ε, και οι αστυνομικέ αρχές στα διάφορα κράτη-μέλη. Δηλαδή πώς ε, ουσιαστικά καταλήγουν στη μεθοδολογία και είναι δύσκολο να καταλήξουν σε καταπολέμηση των οργανώσεων της μαφίας ή των τρομοκρατικών οργανώσεων. Επίσης ε, πρέπει να προσθέσουμε ότι καθώς αυξάνονται αυτά τα φαινόμενα στα διάφορα κράτη-μέλη ε, κρούεται ο κόδωνος του κινδύνου στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν η σχέση μεταξύ ασφαλείας και ελευθερίας είναι πάντοτε μια σχέση που πρέπει να είναι εξισορροπημένη. Θέλω να προσθέσω και κάτι σημαντικό που είναι η προστασία των θυμάτων. Συχνά το θέμα αυτό διαφεύγει ε, και της προσοχής ε, των ευρωπαϊκών πολιτικών. Ε, έχουμε το αυτό το πολύ σοβαρό φαινόμενο της εμπορίας ανθρώπων στα νότια σύνορα της Ευρώπης και έχουμε και τη μετανάστευση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω κάποιον άλλο από τα Εθνικά Κοινοβούλια να θέλει το λόγο. Έτσι λοιπόν θα δώσω το λόγο στο συνάδελφο την κυρία Αναγκόμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μικρόφωνο παρακαλούμε. Sorry. I thought I had. Ε, Ευχαριστώ. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Ράιτ αν ακριβώς ε, στην γνώμη που σύστησε ε, ο καθηγητής, αν η Ευρωπόλα είχε έναν εργό ρόλο στην αξιολόγηση του κόστους του οργανωμένου κλίματος και από την άλλη ο προσδιορισμός στρατηγικών θεμάτων ε, αν ε, ένα από τα θέματα αυτά στη σημερινή συγκυρία μήπως θα πρέπει να είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς και η κατά πολέμηση των tax havens αυτών των φορολογικών παραδείσων ε, και δεν μιλάω μόνο και για υπεράκτης εταιρείε, βρίσκονται και στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και δεν ε, έχουμε μόνο φαινόμενα κάποιων αποστολής κάποιων χρημάτων σε τρίτες χώρες αλλά ουσιαστικά έχουμε και χρησιμοποίηση τέτοιων ποσών των πολιτών και μάλιστα όταν έχουμε τέτοια εποχή κρίσης, αυτό πρέπει να το λάβουμε περισσότερο υπόψη. Αυτό που μας είπε ε, τι κάνει η Ιντερπολ ε, ο κύριος Γουέιν Ράιτ, αλλά δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλές καθυστερήσεις ε, μεταξύ των φορέων και των οργανισμών των δικών μας κρατών μελών. Δυστυχώ αυτέ οι καθυστερήσει έχουν πάρα πολύ αρνητικά αποτελέσματα. Παραδείγματο χάρη έχουμε καθυστέρηση μεταξύ, ε, στη συνεργασία των δικαστικών αρχών μεταξύ Πορτογαλία ε, και Γερμανία. Παραδείγματο χάρη έχουμε την υπόθεση τη πώληση των γερμανικών υποβρυχίων στην Πορτογαλία. Και αυτή η έρευνα καθυστερεί πάρα πολύ. Δεν έχει γίνει μια κοινή έρευνα στην υπόθεση αυτή ε, ε, ε, χρειάστηκαν πάνω από δύο χρόνια, από το 2008, χρειάστηκαν πάνω από το δύο χρόνια για να λάβουν οι δικαστικέ αρχές τα απαραίτητα στοιχεία από τις αρχές τη άλλη χώρα. Έτσι λοιπόν, ο ρόλος εδώ των οργανισμών αυτών σε τέτοιε υποθέσει είναι πάρα πολύ σχετικό. Μάλιστα, ευχαριστώ κύριο Σιμπερτ Μπίκερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε ενώ διάφοροι οργανισμοί τους οποίους έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσαν να κλείσουν χωρίς να αντιλαμβανθούμε καν ότι καταργηθήκανε νομίζω ότι θα υπήρχε κατακραυγή εάν αρχίσαμε να κάνουμε τις ίδιες σκέψεις για την Ευρωπόλη η οποία είναι ένας πρότυπος οργανισμός για ολόκληρο την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για το σχέδιο μη μιας κοινή Ευρώπης και τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά. Ευχαριστώ τον κύριο Wayne Wright και τον συγχαίρω για την εικόνα αυτού του οργανισμού. Χαίρομαι ότι υπάρχει αυτό το μέσο που συμβάλλει στην ασφάλεια στην Ευρώπη και που, για το οποίο μπορούν να, και οι Ευρωπαίοι πολίτες να είναι ήσυχοι ότι τους προστατεύει. Ε, θεωρώ ότι είναι ε, ένα, ε, ε, ένας οργανισμός ο οποίος ελέγχεται ίσως περισσότερο από όλους τους άλλους στην Ευρώπη και γι' αυτό σήμερα και αύριο δεν πρέπει να σκεφτόμαστε πώς μπορούμε να ελέγξουμε περαιτέρω αυτό τον οργανισμό ο οποίος ούτως ή άλλως αναφέρεται σε έναν οργανισμό για την αστυνομική συνεργασία τον οποίο ελέγχουμε ήδη πάρα πολύ. Απλούστατα πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα ε, ε, μέσα ελέγχου που έχουμε για να συμβάλλουμε ε, και να συνδράμουμε το, τη Europol στην καταπολέμηση της οργανωμένης εγκληματικότητας και να μπορέσουμε να πούμε εις την αστυνομία αλλά και και στους πολιτικούς τι μπορεί να επιτύχει η Europol ε, ε, στον τομέα αυτό. Εφόσον έχουμε τόσους ε, εκπροσώπους εμπειρογνώμονες από τα Εθνικά Κοινοβούλια όλων των χωρών γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι ειδικοί αυτοί τι πρέπει να κάνουν τα κράτη-μέλη και γνωρίζουν επιπλέον σε ποιους τομείς η Ευρωπόλ μπορεί να είναι πιο αποδοτική και πού μπορεί να στηριχθεί για να χρησιμοποιήσει την εμπειρία της προς όφελος των πολιτών. Υποθέτω ότι αυτό είναι το νόημα μίας τέτοιας συνεδριάσεως και όχι να σκεφτούμε τι άλλους οργανισμούς θα μπορούσαμε να καταρτήσουμε για να ελέγχουμε την Ευρωπόλη η οποία ελέγχεται ήδη πάρα πολύ. Δεν είναι αυτός ο στόχος ενός τέτοιου θεσμικού οργάνου. ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιος άλλος ε, στην αίθουσα ο οποίος θέλει να κάνει σχόλια. Αν όχι, τότε επανερχόμαστε εις ε, του, τα μέλη ε, του, της Τράπεζα και ξεκινάμε τον κύριο Wainwright της Europol. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, σχετικά με τις ερωτήσεις της κυρίας Σάντα Μαρτίνη. Ήταν ε, πολύ καλές οι παρατηρήσεις που έκανε για την έλλειψη κοινή ερευνητικής ε, κουλτούρας στην Ευρώπη και υπήρχε απουσία μια τέτοια μεθοδολογίας και συνεχίζει να υπάρχει. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια μπόρεσε να βελτιώσει την νομοθεσία και να επιτύχει καλύτερο συντονισμό της αστυνομικής δράσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με το Eurojust και με άλλα μέτρα όπως το Ευρωπαϊκό Ένταρμα Συλλήψεως. Αλλά πέραν αυτού αντιλαμβάνομαι καθημερινά ότι έχουμε πάρα πολλούς αστυνομικούς από πάρα πολλές χώρες που εργάζονται στον οργανισμό μας και ο καθένας έχει τις δικές του ιδέες για το πόσο πρέπει να κάνει μία έρευνα βάσει της εμπειρίας που έχει σε εθνικό επίπεδο. Οπότε ε, πρέπει να πούμε ότι η εφαρμογή που έχει γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο μας βοηθάει πάρα πολύ και μας επιτρέπει να μεταδώσουμε σε όλα τα κράτη-μέλη ένα νέο πρότυπο για την αποτελεσματική αστυνόμευση στην Ευρώπη. Να εντοπίζουμε τις σωστές προτεραιότητες και να εξασφαλίζουμε ότι θα υπάρχει στους τομείς προτεραιότητας η πλέον αποτελεσματική αντιμετώπιση και να υπάρχει και ο συντανισμός ο οποίος θα επιτρέψει στις αστυνομίες των διαφόρων κρατών μελών να καταπολεμήσουν από κοινού και να λύσουν τα προβλήματα τα οποία έχουμε εντοπίσει. Ε, ξέρω ότι η κυρία Χιμένες Μπεχέρο θα επανέλθει στο θέμα αυτό γιατί την ενδιαφέρει ιδιαιτέρως. Όσον αφορά τον κύριο Γκόμες και τον ε, κύριο Μόναρ σχετικά με το κόστος του οργανωμένου εγκλήματος έχει γίνει κάποια συζήτηση για το εάν θα έπρεπε στη φετινή αξιολόγηση των εγκλημάτων να περιληφθεί και αυτό το στοιχείο. Τελικά όμως ε, αποφασίσαμε να μην το περιλάβουμε διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να εκφράσουμε ποσοστιαία το κόστος. Υπάρχουν ε, διάφορα στοιχεία τα οποία γνωρίζουμε και μπορούμε να κοστολογήσουμε όπως το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και έχουμε εντοπίσει και ορισμένους άλλους τομείς. Αλλά νομίζω ότι οι υπολογισμοί αυτοί δεν θα αντέξουν σε προσεκτική ε, εξέταση γιατί δεν πρέπει κανείς να αναφέρεται μόνο στις, ε, στο άμεσο κόστος αλλά και στο έμεσος όλα τα ε, θύματα παραδείγματος χάρη ε, της, ε, του εμπορίου ναρκωτικών. Ε, Ένα άλλος τρόπος με τον οποίο το οργανωμένο έγκλημα οδηγεί σε κοινωνικές εντάσεις μέσα σε κοινωνίες, πώς επηρεάζει τις διάφορες κοινωνίες και τους πολίτες. Έχουμε δηλαδή διάφορους τομείς στους οποίους ο κύριος Μόναρ και η συνάδελφοι συνάδελφοί τους θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν. Όσον αφορά τη διαφθορά, και την καταπολέμησή της. Πρέπει να ε, συμφωνήσω ότι αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα ε, που αντιμετωπίζουμε από το οργανωμένο έγκλημα διότι το διαπιστώνουμε όχι μόνο διεθνώς αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να εφαρμόσουμε παραδείγματος χάρη μέτρα κατά πολέμησης του ξεπλήματος ε, μαύρου χρήματος και ε, πρέπει ε, να σας πω ότι πιστεύω ότι η Europol μπορεί να βελτιωθεί στον τομέα αυτό εάν υπάρχει καλύτερος συντονισμός και τέλος ε, κύριε Πίρκερ σας ευχαριστώ για τις ε, παρατηρήσεις σας και για την ερώτηση για το μέλλον. Δεν είναι ότι χρειαζόμαστε περισσότερο έλεγχο αλλά πιο αποτελεσματικό τρόπο εξασκήσεως αυτού του ελέγχου και επίσης εποπτεία από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ε, δεν είναι μόνο το θέμα όπως σας είπα να υπάρξει ένας δημοκρατικός τρόπος ε, εποπτείας έχουμε τις δυνατότητες αυτές μπορούμε να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα και στο μέλλον και έχουμε δυνατότητες και για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο που είναι ε, ε, μια πραγματική πρόκληση στον τομέα μας. Η κυρία Χιμένες, μάλιστα. Θέλω να απαντήσω στον κύριο Σαντεμαρτίνο ο οποίος ε, είπε ότι χρειάζεται περισσότερη νομοθεσία και πρέπει να υπάρχει περισσότερη προσοχή ως προς τα θύματα. Συμφωνώ με όσα είπατε και εγώ όταν έφτασα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχα αυτή την εντύπωση ότι δηλαδή χρειαζόταν να νομοθετήσουμε περαιτέρω και ότι η ζυγαριά έγινε περισσότερο προς την πλευρά του δράστη παρά προς την πλευρά των θυμάτων. Και πρέπει να σας πω ότι θα εγκρίνουμε τώρα στην Ολομέλεια τον επόμενο μήνα. Ήταν κάπως δύσκολη η πορεία, αλλά μετά από ένα χρόνο μπορούμε να πούμε ότι έχουμε αυτή την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας πλέον. Πρόκειται για μια εντολή προστασίας των θυμάτων αυτό σημαίνει ότι αν ένα άτομο έχει εκδοθεί εντολή απομάκρυνση, μάλλον συγγνώμη, αν ένα άτομο έχει μια εντολή απομάκρυνσης ε, ενό ατόμου που συνιστά απειλή και μπορεί να ταξιδέψει το άτομο αυτό, να μεταβεί σε άλλη χώρα και να την χάνει τη ίδια προστασία, χωρί να ξεκινήσει μια διαδικασία για την προστασία των θυμάτων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα βοηθήσει όλα τα θυμάτα οικογενειακή βία αλλά και οποιοδήποτε άλλο θύμα το οποίο ε, γνωρίζει το άτομο που το απειλεί. Υπήρξε πολύ μεγάλη έλλειψη ε, για την προστασία των θυμάτων και έτσι λοιπόν η Κομισιόν αποφάσισε να υιοθετήσει ένα πακέτο για τα θύματα και τώρα θα έχουμε ένα αντεμήνυμις πακέτο μέτρων για τα θύματα και θα ε, χρησιμεύσει για όλα τα θύματα και θα ισχύει σε όλες τις χώρες από την Βουλγαρία ως την Ισπανία και θα καλύπτει όλα τα θύματα με ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες ομάδες και μιλάμε για τους ανηλίκους, ε, θύματα τρομοκρατίας, θύματα εμπορίας ανθρώπων. Λαμβάνουμε πάρα πολλές πληροφορίες ε, και Καλό τα εθνικά κοινοβούλια να μας στείλουν ε, κάθε συνεισφορά αν, θέλουμε να, αν θέλουν ε, να συνεισφέρουν και να προσθέσουμε κάτι σε αυτή τη σημαντική νομοθεσία. Μάλιστα, ευχαριστώ. Επανερχόμαστε στον ε, καθηγητή Μόναρ. Ευχαριστώ. Σας κατευχαριστώ. Θα ήθελα απλώς να κάνω μερικά πρόσθετα σχόλια για αυτό το θέμα της διαφοροποίησης και των διαφορών μάλλον μεταξύ των ηθών που υπάρχουν στις αστυνομικές υπηρεσίες. Παραμένει πρόβλημα γιατί δημιουργεί παρεξηγήσεις και εμποδίζει την αστυνομική συνεργασία. Βέβαια εδώ πρέπει να γνωρίζουμε ότι το θέμα είναι λίγο πιο μακροπρόθεσμο. Δεν μπορούμε να εναρμονίσουμε ήθη και πολιτισμούς ακόμη και αν είμαστε διευθυντέ της Europol. Δεν γίνεται αυτό με νομοθεσία δηλαδή έστω και ενωσιακή. Ο Φερνάν Μπροντέλ είχε πει κάποτε ότι οι νοοτροπίες είναι φυλακές μακράς διαρκείας. Είναι λοιπόν πρόβλημα, αλλά η Ευρώπη νομίζω παίζει πολύ επικοδομητικό ρόλο εδώ, γιατί φέρνει σε συνεργασία αξιωματούχους αστυνομιών. Μπορεί μεν να είχαν αντιδράσει αλλιώς αν ανήκαν σε άλλο κράτος μέλος, αλλά τουλάχιστον πληροφορούνται. Νομίζω λοιπόν ότι ο ρόλος της Ευρωπόλ είναι ουσιαστικός και το σημαντικότερο απ' όλα είναι η συνεργασία σε πολύπλευρο επίπεδο μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων. Δεν θεωρούμε ότι αυτό είναι ασύμβατο με τον αυξανόμενο ρόλο της Ευρωπόλ. Χρειάζεται να συνεχιστεί αυτή η πολύπλευρη αστυνομική συνεργασία πέρα από τα σύνορα της κάθε χώρας. Τώρα για την αξιολόγηση των, της σημασίας των εγκλημάτων Νομίζουμε ότι η Ευρωπόλ δεν έχει ακόμη καταφέρει να δημιουργήσει την κατάλληλη μεθοδολογία για ενιαία αντιμετώπιση γιατί δεν έχει και αρκετούς πόρους, βασίζεται σε εμπειρικά στοιχεία δεν έχει δημιουργήσει καμία ενιαία θεωρία. Εσείς το Ευρωκοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια θα μπορούσατε να υποστηρίξετε την ιδέα η Ευρωπόλ να έχει μια κάποια μεγαλύτερη προτεραιότητα γιατί υπάρχουν χρήματα για την ανάληψη μελετών άρα θα μπορούσε και η Ευρωπόλ να παίζει κάποιο ρόλο όχι ίσως τελικό ή καθοριστικό αλλά να παίζει κάποιο ρόλο και η ίδια ως προς τον καθορισμό των κοντιλίων που χορηγούνται για την ανάληψη ερευνών. Βέβαια όντως είναι και αυτό ένα θέμα αποτελεσματικότερης χρησιμοποίησης των χρημάτων του φορολογούμενου και της φορολογούμενης. Ε, όσο για τα θέματα της διαφθοράς, ναι, συνεχίζει να είναι ένα πολύ λεπτό θέμα και σοβαρό γιατί όλοι γνωρίζουν ότι χωρίς να πω ονόματα εδώ χωρών υπάρχει σε πολλές χώρες, σε μερικές χώρες μέλη μεγαλύτερο πρόβλημα διαφθοράς από ό,τι σε άλλες και το θέμα είναι πολιτικά ευαίσθητο. Αν έχει στεναρότερη εντολή η Europol ίσως, δεν λέω σίγουρα, ίσως να μπορούσε να αντιμετωπίσει και το πρόβλημα αυτό. η Ένωση έχει προοδεύσει στο θέμα της διαφθοράς, έχει ένα κοινό νομικό υπόβαθρο, μινιμαλιστικό βέβαια, αλλά υπάρχει κάποια πρόοδος. Πρόοδος αργή, αλλά αληθινή. Και αυτό είναι θετικό. Για τους φορολογικούς αραδίσους. Αυτό είναι θέμα που αφορά αποκλειστικά τα κράτη-μέλη. Αν το Συμβούλιο δεχτεί να γίνει κάτι για την καταπολέμησή τους θα γίνει. Αλλά θα έλεγα ότι λόγω των συγκεκριμένων προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε στους εθνικούς προϋπολογισμούς μάλλον ήρθε η ώρα να καταργηθούν, να καταπολεμηθούν οι φορολογικοί παράδεισοι γιατί αυτό θα ωφελούσε πολύ την καταπολέμηση του εγκλήματος. Τέλος, κάτι ίσως επικίνδυνο να το πει κανείς, όταν διαβάζω τις εκθέσεις της Ευρωπόλ καταλαβαίνω ότι πρέπει να ξέρουν πολλά περισσότερα από όσα λένε, δηλαδή ξέρουν ποια κράτη-μέλη δεν συνεργάζονται πλήρως, ενώ η γλώσσα την οποία χρησιμοποιούν είναι πολύ διπλωματική με φημισμούς. Νομίζω ότι εδώ θα μπορούσαν να ονοματίζουν κάπως περισσότερο naming and shaming τους υπεύθυνους. Πριν από μερικούς μήνες ένα άρθρο του Μάριου Μόντι εμφανίστηκε στους Financial Times που έλεγε ότι μέρος του προβλήματος των κρατικών χρεών είναι η υπερβολική ευγένεια που χρησιμοποιείται στην Ένωση. Και νομίζω ότι αυτό ισχύει και σε άλλους τομείς στον τομέα της επιβολής του νόμου επίσης ισχύει. Πρέπει κανείς βέβαια να εκφράζεται διπλωματικά, αλλά τουλάχιστον από ακαδηματικής απόψεως θα έλεγα ότι αν είναι και πιο συγκεκριμένα τα πράγματα, τα φίκα, σίκα και τις κάφη, σκάφη δεν θα ήταν κακό. Α, μάλιστα. Δυστυχώς, πάλι καθυστερούμε. Φτάνουμε στον τελευταίο γύρο τώρα. Τα μέλη του παρακαλώ, όπως ο κύριος Αλέκος Γουίλιαμς, η κυρία Ρενάτε Βέμπερ, ο κύριος Διογέρζη Μόντακ δυστυχώς δεν μπόρεσε να έρθει στα Βρυξέλλας είναι μέλος του Bundestag. Και ο κύριος Ανρί Λαμπέιλ από το Πανεπιστήμιο της Βαγιώνης θα μας τα πει πιο ακαδημαϊκά. Ευχαριστούμε τους προηγούμενους ομιλητές και ομιλήτριες και συνεχίζουμε χωρίς καμία διακοπή στο επόμενο θέμα. Μπορώ να έχω την προσοχή σας παρακαλώ. Λοιπόν, να χρησιμοποιήσουμε καλά το χρόνο μας για να προχωρήσουμε χωρίς χρονοτριβή στο επόμενο σημείο. Καταρχήν, κάνουμε εδώ μια συζήτηση για την οικοδόμηση ενός ευρωπαϊκού δικαστικού χώρου και πώς συνδέεται με τους εθνικούς δικαστικούς χώρους και συγκεκριμένα το ρόλο της Eurojust. Καλωσορίζουμε τον πρόεδρο του σώματος της Eurojust, τον κύριο Άλεντ Βίλιαμ, ο οποίος θα πάρει πρώτο το λόγο. Κύριε Βίλιαμς. Um, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Σας παρακαλώ λέει ο Πρόεδρος αν θέλετε να αποχωρήσετε από την αίθουσα, σας παρακαλώ χωρίς να μιλάτε. Έτσι ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν οι υπόλοιποι την παρουσίαση του κυρίου Williams. Um, Έχουμε μια κρουσία στα αγγλικά ότι ψηφίζει κάποιος με τα πόδια του. Αλλά δεν θα με ακρηγορήσω πάνω από 10 λεπτά. Σας το υπόσχομαι. Σε ό,τι αφορά την εισαγωγή αυτή στο θέμα. Αυτό που δεν πρόκειται να κάνω είναι να αντικατοπτρίσω την ε, πολύ γλαφυρή ε, παρουσίαση του κυρίου Wainwright σε σχέση με τον αριθμό ε, των ελέγχων που υπάρχουν και σε ό,τι αφορά τη Europol και σε ό,τι αφορά τη Eurojust ως προς την δημοκρατική λογοδοσία. Υπάρχει φυσικά μια διαφορά μεταξύ της προσέγγισης που ακολουθείται υπό τη συνθήκη της Λισαβόνας απέναντι στη Eurojust και στη Europol. Η Europol ε, υπόκειται σε ελεγχό και η Eurojust, σύμφωνα με τη συνθήκη, υπόκειται σε αξιολόγηση. Και ο έλεγχος ε, σκρούτινη ακούγεται κάπως ε, πιο αυστηρό από την αξιολόγηση. Τώρα, εγώ θα προσπαθήσω να απαντήσω συντομία σε δύο ερωτήματα που ελπίζω θα αποτελέσουν ένα είδος εισαγωγής στο έργο της Eurojust. Το πρώτο ερώτημα έχει να κάνει σε σχέση με το ότι είδους ε, λογοδοσία θα πρέπει να εφαρμόζεται να ισχύει για έναν οργανισμό όπως η Eurojust που στην προηγούμενη συνθήκη περιγραφόταν ως ε, μονάδα δικαστικής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι είναι εύκολο να πούμε σχετικά γρήγορα τι είδου λογοδοσία δεν θα πρέπει να εξετάζεται εδώ από το Ευρωπαϊκό και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Και αυτό είναι η επιχειρησιακή λογοδοσία. Εδώ ε, βασίζομαι σε μια πολύ χρήσιμη έκθεση που προήρθε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο των Οργανισμών Ασφαλείας και Πληροφοριών της Ευρωπαϊκή Ένωση που αναφέρθηκε νωρίτερα σήμερα το απόγευμα από την κυρία Μπερσολίνου. Γιατί δεν ε, είναι σκόπιμο να ε, έχουμε λογοδοσία σε σχέση με τα επιχειρησιακά ζητήματα ως προς τη Eurojust η απάντηση είναι αρκετά απλή. Αν ε, κάποιος ε, δει ποια είναι η αποστολή της Eurojust, έτσι όπως περιγράφεται στη Συνδίκη της Λισαβόνας, η αποστολή τη είναι να υποστηρίξει και να ενισχύσει το συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών ερευνητικών και εισαγγελικών αρχών βάσει πληροφοριών που προέρχονται από αυτές τις αρχές και από την Europol. Έτσι λοιπόν η Eurojust ουσιαστικά υπάρχει προκειμένου να συντονίζει τις προσπάθειες των ευρωπαϊκών οργανισμών όπως Europol, Frontex και Olaf αλλά επίσης και να συνεργάζεται πολύ στενά με τις εθνικές ερευνητικές και διοικητικές αρχές και εισαγγελικές αρχές, με συγχωρείτε. Δεύτερον, για να στραφώ στο θέμα της διεπαφής μεταξύ Eurojust και εθνικών, ερευνητικών και εισαγγελικών αρχών. Είναι υβριδικός φορέας η Eurojust, δηλαδή αποτελείται από εισαγγελείς, δικαστές και αστυνομικούς από τα κράτη-μέλη, αλλά και από άτομα που διορίζονται απευθεία από την Κομισιόν ουσιαστικά, από τις Βρυξέλλες. Ε, σε ό,τι αφορά την κατανομή σε αριθμούς, η Eurojust είναι ένας μικρός ελπίζω αποτελεσματικός οργανισμός. Έχουμε περίπου 45 εισαγγελείς ε, από τα κράτη-μέλη που εργάζονται στην Eurojust και πληρώνονται από τα κράτη-μέλη σε στενή συνεργασία με τις αρχές των κρατών μελών. Έχουμε περίπου 200 απασχολούμενους ε, από την Κομισιόν, από ε, τον τομέα της Eurojust, ε, τομέα προπολογισμού της Eurojust και έχουμε και κάτι πολύ χρήσιμο για την οικοδόμηση ενός χώρου δικαιοσύνης ασφάλειας έχουμε και τους αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες. Ε, περίπου 15 έχουμε στη Eurojust, προέρχονται από τα κράτη-μέλη, εργάζονται στη Eurojust σε συγκεκριμένες επιχειρησιακές περιπτώσεις και κατόπιν επιστρέφουν στα κράτη-μέλη για να γνωστοποιήσουν ε, πώς εξιέχει τον εργαζόμαστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να καταπολεμούμε το οργανωμένο έγκλημα. Ελπίζω να σας δώσω ένα, ένα καλό παράδειγμα. Σκεφτείτε μια περίπτωση όπου οι αστυνομικές αρχές ε, ενός κράτους μέλους ε, στέλνει πληροφορίες του Europol κατόπιν σύλληψης ενός ε, εμπόρου ναρκωτικών. τους χάρη λαμβάνονται πληροφορίες από αυτόν σχετικά με τα, με τα νούμερα, τα τηλεφωνικά που βρήκαν στο τηλέφωνο του ανθρώπου αυτού κατόπιν στέλνονται αυτά τα στοιχεία στη Europol, εξετάζονται σε ένα από τα αρχεία δεδομένων εργασία προ ανάλυση, τα analysis work files και επίση προκύπτει από αυτό ότι ο άνθρωπο αυτό ήταν, ε, είχε έρθει σε επαφή με άλλους εμπόρους ε, ναρκωτικών σε άλλα κράτη-μέλη. Πρόκειται για μια επιχείρηση η οποία υλοποιείται προδραστικά. Υπάρχουν αποδείξεις ότι υπάρχει μια κλιματική οργάνωση η οποία δραστηριοποιείται και γίνεται προφανές ότι προκειμένου να παρακολουθούν διάφορα τηλέφωνα είναι απαραίτητο να υπάρχουν ε, άδειε δικαστική ε, άδεια σε ορισμενα κρατημέλη κράτη-μέλη. Και κάτι τέτοιο δεν είναι πάντοτε εύκολο επειδή υπάρχει διαφορο... υπάρχουν διαφορές ε, στην νομοθεσία μεταξύ των κρατών μελών και σε μετέπειτα στάδια θα είναι απαραίτητο να διασφαλίσουμε ότι οι τραπεζικοί λογαριασμοί των εμπόρων ναρκωτικών σε αυτή την εγκληματική ομάδα έχουν δεσμευτεί. Μπορεί να ισχύουν διάφοροι κανόνε σε ό,τι αφορά το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων σε ένα κράτο μέλο σε σχέση με ένα άλλο και θα υπάρχει αναγκαιότητα έκδοση Ευρωπαϊκού Εντάλματο Σύλληψη και πάλι έχουμε δικαστικέ πράξει στα περισσότερα κράτη-μέλη. Έτσι λοιπόν η Eurojust εμπλέκεται σε στενή συνεργασία με τη Europol ως αποτέλεσμα αυτής της αρχικής επαφής. Εδώ, κατά κάποιο τρόπο, για να σας ε, το πω πάρα πολύ σύντομα, έχετε ένα παράδειγμα για το πώς πρέπει να εργάζονται τα πράγματα, συγγνώμη, πώς πρέπει να λειτουργούν τα πράγματα σε ό,τι αφορά στη Eurojust. Και τελικά τι συμβαίνει όταν προχωρούν οι επιχειρήσεις με το συντονισμό της Eurojust και έχουμε περίπου 150 συνεδριάσεις συντονιστικές στη διάρκεια ενός έτους σε τέτοιες περιπτώσεις. Ο πραγματικός δικαστικός έλεγχος που ασκείται ως προς τη χρήση των πληροφοριών, ως προς το συντονισμό αυτών ε, των ε, δράσεων ε, που λαμβάνονται κατά των εγκληματιών, όλα αυτά υπόκειται σε εθνικό δικαστικό έλεγχο. Και γι' αυτό θα έλεγα εγώ ουσιαστικά ότι η δημοκρατική λογοδοσία της Eurojust δεν θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνει το επιχειρησιακό σκέλος, την επιχειρησιακή δουλειά που κάνουμε. Το μόνο ε, που θα πω για να διαφοροποιηθώ είναι ότι ε, στο βαθμό που Eurojust ε, μάλλον υπάρχουν όπως και σε άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς έτσι και στην Eurojust κάποιες προτεραιότητες που από τα εθνικά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλια εμείς εργαζόμαστε βάσει των προτεραιοτήτων που έχουν χαραχθεί για μας από τα αρμόδια όργανα εδώ στις Βρυξέλλες, φυσικά και με τη συνεισφορά των νομοθετών. Συγκεκριμένα έχω κατά νου το έργο που γίνεται από την Κόζη και την απέτηση δυνάμει του άρθρου 71 ότι πρέπει να υπάρχει ενημέρωση των εθνικών και, των εθνικών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως προς τις δραστηριότητες αυτές. Έτσι λοιπόν, κατά κάποιο τρόπο, αυτή είναι οι κανόνες που ισχύουν για την Eurojust. Καλωσορίζουμε την δημοκρατική λογοδοσία σε όλες τις δραστηριότητές μας, αλλά σε ό,τι αφορά το επιχειρησιακό μας έργο, για τους λόγους που σας παρουσίασα και νομίζω ότι και η πλειοψηφία των νομοθετών συμφωνεί, Δηλαδή ε, δεν θα ήταν ε, σκόπιμο να γίνεται έλεγχος της ε, επιχειρησιακής δουλειάς των λεπτομεριών αυτή τη επιχειρησιακή δουλειά. Πώ μπορούμε να βελτιώσουμε όμω το έργο τη Eurojust και ω προ το επιχειρησιακό αντίκτυπο και ω προ τη λογοδοσία. Εδώ έχω μία δική έκκληση να απευθύνω. Θα έλεγα καταρχήν ότι είναι ζωτική σημασία τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιούν πλήρως το σημερινό διαθέσιμο πλαίσιο ως, ε, σε ό,τι αφορά τη Eurojust συγκεκριμένα η Eurojust δυνάμει της νέας απόφασης από τις 4 Ιουνίου φέτος, δηλαδή μόλις πριν δύο μήνες υιοθετήθηκε ε, έχει τεθεί υποχρέωση στα κράτη-μέλη να παρέχουν στη Eurojust ε, λεπτομερή στοιχεία σε σχέση με οποιαδήποτε υπόθεση ε, σοβαρή διασυνοριακού εγκλήματος. Έτσι λοιπόν, οποιαδήποτε τέτοια σοβαρή περίπτωση θα πρέπει να κοινοποιείται στη Eurojust. Έχουμε επίσης ε, δημιουργήσει και τις κοινέ ερευνητικέ ομάδες, σίγουρα θα τις έχετε ακούσει και δυνάμει της νέας ε, απόφασης προωθούμε το εθνικά συστήματα συντονισμού της Eurojust, δηλαδή η εικονικά γραφεία για την Eurojust σε κάθε ένα από τα κράτη-μέλη. Αλλά σε ένα ευρύτερο επίπεδο νομίζω ότι είναι επίσης πολύ σημαντικό και θίγει τη δημοκρατική λογοδοσία και ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα Εθνικά Κοινοβούλια είναι ε, η ανάληψη νομοθετικών ε, μέτρων. Εδώ έχω κατά νου όχι μόνο το άρθρο 85 και το άρθρο 86 της Συνθήκης της Λισαβόνας, που θα αναφέρω στη συνέχεια, αλλά και πολύ συγκεκριμένα μέτρα που θα φτάσουν σύντομα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σκέφτομαι την Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνα που θα φέρει μία επανάσταση σε ό,τι αφορά ε, την ε, διασυνορία και συνεργασία σε ποινικέ υποθέσει. Ε, θα αντικατασταθεί ένα παρχαιωμένο σύστημα την εργασία των κρατών μελών ε, σε ό,τι αφορά τις ε, διασυνοριακές ποινικέ έρευνες. Υποθέτω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εξετάσει θετικά την πρόταση για αυτή την Ευρωπαϊκή Ερευνητική Εντολή. Θα πρόκειται για ένα μέσο που θα προσφέρει και στους αγγελείς και στις ε, διοκτικές αρχές τη δυνατότητα να συνεργαστούν αποτελεσματικά μέσω ενός νέου μέσου αναγνώρισης. Να συνεργαστούν λοιπόν αποτελεσματικά μεταξύ τους. Και το αναφέρω αυτό για ένα λόγο και αυτό έχει να κάνει με την αναλογικότητα. Όταν αυτό το μέσο έλθει εδώ για εξέταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όταν θα εξεταστεί και από τα Εθνικά Κοινοβούλια, ε, υπάρχει ένα μειονάκτημα με τη γενική ε, εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης ότι δεν εφαρμόζεται παρκώς η αρχή της αναλογικότητας. Αν οι νομοθέτες μπορούν να διασφαλίσουν ότι η αρχή της αναλογικότητας αντικατοπτρίζεται ορθά στη νέα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα προς τα μπρος για την καταπολέμηση του διασυνεωρικού οργανωμένου κλίματος. Έχω και κατά νου το χρόνο. Ανέφερα και το άρθρο 85 και το πρόταση κανονισμού που θα καταταθεί πιθανότατα το φθινόπωρο του 2012. Δυνάμει το άρθρο 85 υπάρχουν ε, δύο τρόποι που μπορεί να μεταρρυθμιστεί η Eurojust για να είναι πιο αποτελεσματική για το μέλλον. Υπάρχουν διατάξεις στο άρθρο 85 που έχουν να κάνουν με την επέκταση των αρμοδιοτήτων της Eurojust. Ουσιαστικά δυνατότητα κίνησης ερευνών και έναρξη ερευνών και δυνατότητα ε, να επιλύσει συγκρούσεις δικαιοδοσίας ε, αυτό το θέμα των αρμοδιοτήτων δεν θα αντικατοπτριστεί πιθανόν σε μια απόφαση σε μια πρόταση κανονισμού για τη Eurojust. Αυτό που πρέπει να ρυθμιστεί και να σκεφτούν οι νομοθέτε είναι η ίδια και η διαχείριση τη Eurojust, η διακυβέρνηση τη Eurojust. Και φυσικά δυνάμει τη διαδικασία στην απόφαση δίνεται η δυνατότητα έτσι για άμεσο δημοκρατικό έλεγχο σε ό,τι αφορά την πολιτική διαχείριση και τη χρηματοδότηση της Eurojust. Συγγνώμη, έχω υπερβεί το χρόνο. Θέλω να αναφερθώ όμω και στο άρθρο 86 και στη δυνατότητα να έχουμε ένα ε, γραφείο δημοσίου κατηγορού. Αυτό είναι ένα πολύ λεπτό και πολύ πλοκό θέμα και αν μπορώ θα ήθελα να το παρακάμψω και να αναφερθώ και πάλι στις διατάξεις, στις εφιστάμενες διατάξεις και στην αφαιρμένη απόφαση Eurojust. Απαιτείται από τα κράτη-μέλη να παρέχουν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις στη Eurojust πληροφορίες για οποιαδήποτε διασυνορική υπόθεση που ε, ερευνούν ε, και έχει να κάνει με επίθεση σε κάποιο οικονομικό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Eurojust θα είναι σε θέση από τη σκοπιά των αποδείξεων να παράσχει χρήσιμες πληροφορίες για τους νομοθέτες όταν θα εξετάσουν αυτή τη συγκεκριμένη πτυχή. Σας ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ τον κύριο Williams για αυτή την ε, διεξοδική παρουσίαση ε, του, ε, του σώματος της Eurojust και τώρα δίνω το λόγο στην εισηγήτρια σχετικά με το Eurojust την κυρία Ρενάτε Βέμπερ μέλος Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών και ε, η συγγήτρια για το θέμα της επιλογής ε, της ε, δικαιοδοσίας σε περίπτωση ποινική προσφυγής. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, χαίρομαι που είμαι εδώ σήμερα όπως και πριν από ένα χρόνο όταν είχαμε κάνει τη συνεδρίαση με τα Εθνικά Κοινοβούλια επειδή στηρίζω πάρα πολύ αυτές τις συνεδριάσεις και τη στενότερη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων. Θα ε, ε, θα ξεκινήσω από εκεί που σταμάτησε ο πρόεδρος Βίλιαμς διότι στην αρχή ανέφερε ότι σύντομα ε, ελπίζουμε ότι θα έχουμε νομοθετικές αλλαγές. Δεν νομίζω ότι θα είναι και τόσο σύντομα αλλά έχουμε κάποιο χρόνο να ετοιμαστούμε και να αντιληφθούμε τι επιζητούμε με αυτή τη νέα νομοθεσία. Και αυτό θα μας βοηθήσει πολύ. Όπως μας βοήθησε και θα συνεχίσει να μας βοηθά το να καταρτίζουμε τη μελέτη αυτή ε, την ε, οποία ε, λάβαμε την περασμένη εβδομάδα και σας τη συνιστώ να τη διαβάσετε τη λάβαμε όπως είπα την περασμένη εβδομάδα στην Επιτροπή Ελευθεριών πρόκειται για μια ανεξάρτητη μελέτη εμπειρογνωμόνων από κάποια ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και θα ήθελα να συζητήσουμε ορισμένα από τα θέματα που πραγματευόταν διότι είναι σχετικά με αυτά τα οποία συζητάμε σήμερα. Ε, είπε ο πρόεδρος Βίλιαμ ότι θα έπρεπε ε, να ε, συμμετέχουμε στη δημοκρατική λογοδοσία. Πρέπει λοιπόν σαν επόπτες έχοντας μία εντολή επόπτη των ευρωπαϊκών εργανισμών στον τομέα αυτό ποιος είναι ο στόχος μας. Μιλάμε για εποπτεία της πολιτικής, της διοίκησης, των οικονομικών και δεν νομίζω ότι αυτά τα θέματα είναι ε, φιλεγόμενα. Βεβαίως έχουμε και νομοθετική ε, ε, εντολή αλλά το καλύτερο είναι να συζητάμε με το Συμβούλιο της Eurojust και να δούμε τι άλλους τομείς πολιτικής ενδέχεται να χρειάζεται να προωθήσουν. Όσον αφορά τα οικονομικά οικονομικά και την διοίκηση. Έχουμε την Επιτροπή προϋπολογισμού, την Επιτροπή Ελευθεριών που μπορεί να συμβάλλει στην κατάρτιση του προϋπολογισμού. Έχουμε την ε, Επιτροπή ε, Ελέγχου του Προϋπολογισμού, δηλαδή είμαστε καλά κατεπτυσμένοι διότι ο έλεγχος αυτός είναι πολύ αυστηρός και βλέπουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να εμπλακεί εις ε, το Διοικητικό Συμβούλιο και να εκπροσωπείται ούτε μπορεί να ε, εμπλακεί εις ε, τον καθορισμό του Προέδρου ή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για να μείνει ουδέτερο το Κοινοβούλιο και να είναι πιο αποτελεσματικό όταν εξασκεί την ε, εντολή εποπτείας. Βέβαια αυτό όπως αντιλαμβάνετε είναι κάτι το οποίο συζητείται και αμφισβητείται σε αυτό το κοινοβούλιο γιατί θα θέλαμε να μπορούμε τουλάχιστον να επηρεάζουμε την ε, επιλογή του Πρόεδρου αλλά θα το ξανασκεφτούμε. Η αλήθεια όμως είναι <clears throat> ότι το πιο ευαίσθητο θέμα όταν μιλάμε για την εποπτεία είναι η ε, συγκέντρωση των ε, πληροφοριών από την Eurojust, από την Europol και από τη Frontex τι πληροφορίες πρέπει να λαμβάνουμε ή τι δικαιούμαστε να λαμβάνουμε διότι η πρώτη σύσταση της μελέτης αυτής ε, λέγει και το αναφέρω ότι είναι βασικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξασφαλίσει ότι οποιαδήποτε ε, νέα ρύθμιση για την εποπτεία αυτών των οργανισμών δεν θα αποτρέψει ε, τα κράτη-μέλη από το να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πλατφόρμες συνεργασίας. Δηλαδή, εάν είστε πολύ απαιτητικοί από τους οργανισμούς αυτούς, τους επιβαρύνετε πάρα πολύ, τότε τα κράτη-μέλη θα αποστραφούν, θα προτιμήσουν τη διμερή συνεργασία αντί να χρησιμοποιήσουν την Eurojust ή την Europol. Αλλά, βέβαια, από την άλλη πλευρά δικαιούμαστε να λάβουμε πληροφορίες και πρέπει να δούμε πώς θα τα συνδυάσουμε αυτά τα δύο θέματα. Και ίσως ή μάλλον με τα βεβαιότητος, πιστεύω ότι αυτό είναι σημαντικό για την επίλυση των προβλημάτων, πρέπει όταν κοιτάζουμε τι πληροφορίες χρειαζόμαστε να γνωρίζουμε ότι λαμβάνουν πληροφορίες και από τα κράτη-μέλη και από διάφορα εθνι... και διάφορους εθνικούς οργανισμούς ε, την ε, αστυνομία, τα δικαστήρια, αλλά πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στα εθνικά κοινοβούλια και στους εθνικούς οργανισμούς να παρακολουθούν και να εποπτεύουν σε εθνικό επίπεδο τις εργασίες. Και γι' αυτό θα πρέπει να γνωριζόμαστε καλύτερα και να συνεργαστούμε περισσότερο, διότι διαφορετικά ε, θα υπάρχουν επικαλύψεις με το ότι γίνεται ήδη σε εθνικό επίπεδο. Μια άλλη δυνατότητα είναι να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο, όχι όπως τώρα που είναι πολύ περιορισμένη η συνεργασία αλλά να μπορέσουμε να συνεργαστούμε καλύτερα με τις, ε, τους κοινού εποπτικούς οργανισμούς διότι εμείς σαν Ευρωπαίοι έχουμε καταρτήσει αυτούς τους οργανισμούς με συγκεκριμένη εντολή να ε, εξασκούν μία πολύ αυστηρή εποπτεία στους οργανισμούς αρφούς οπότε πρέπει να τους έχουμε από δίπλα ε, διότι μέσω αυτών ουσιαστικά έχουμε δικαίωμα να εξετάσουμε όλα τα στοιχεία, όλους τους φακέλους και στη συνέχεια αυτοί θα έρθουν και θα μας ενημερώσουν αν κάτι πήγε στραβά. Και αν πήγε στραβά να, θα ζητήσουν από τις οργανώσεις να ε, διορθώσουν αυτά που έχουν γίνει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό που κάνει το Κοινοβούλιο είναι απλώς να συναντάτε με τους εποπτικούς οργανισμούς μόνο όταν ε, καταρτίζεται η εθνική η ετήσια έκθεση και δεν επαρκεί. Πρέπει επίσης να σας πω ότι η μελέτη αυτή είναι πολύ σαφής και λέγει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν πρέπει ε, να έχει πρόσβαση εις ε, τις βάσεις δεδομένων ε, των πολιτών κρατών μελών ή τρίτων κρατών γιατί θα παρισφρήσει σε τομείς που δεν είναι της αρμοδιότητός τους και είναι σαφές αυτό διότι πολλές φορές μπορεί να, να έχουμε κάποιο σοβαρό λόγο δηλαδή εγώ προέρχομαι ε, από μία ομάδα η οποία αμφισβητεί ε, την ε, ανάγκη ορισμένων νομοθεσιών θα σας έλεγα όμως ότι αν δεν έχω αρκετή πληροφόρηση πώς είναι δυνατόν να κάνω μία σωστή εκτίμηση του τι γίνεται σε αυτούς τους οργανισμούς και γι' αυτό επανέρχομαι στην ίδια μελέτη η οποία λέγει ότι η πληροφόρηση είναι το οξυγόνο το οποίο τροφοδοτεί την επιποπτεία και πρέπει πάντοτε να υπάρχει δυνατότητα ε, να έχει κανείς ε, ε, τη δυνατότητα να εξετάσει ό,τι είναι σχετικό. Και αυτό αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη, διότι διαφορετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τα δυσκολίας θα γνωρίζει αν πρέπει να αλλάξει την νομοθεσία, εάν πρέπει να κινήσει περισσότερους δημοσιονομικούς πόρους ή αν χρειάζεται άλλων ειδών συνεργασίες. Πώς λοιπόν θα συγκεντρώσουμε αυτές τις πληροφορίες εδώ και πάλι υπάρχει μια συζήτηση πολύ ε, ζωντανή σε αυτό το κοινοβούλιο γιατί έχει συζητηθεί να καταρτιστεί κάποια υποεπιτροπή η οποία θα ασχολείται μόνο με τις διαβαθμισμένες πληροφορίες. Δεν συμφωνούν όμως όλοι με αυτή την ιδέα και ορισμένοι από τους συναδέλφους μας μας λένε ε, όχι η ενημέρωση πρέπει να είναι δημόσια και ανοιχτή και πρέπει να είμαστε λογικοί για το ότι ζητάμε. Γενικώ όμως χρειαζόμαστε ένα μηχανισμό ο οποίος θα επιτρέψει στους ευρωβουλευτές να έχουν πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες. Καταλήγω λοιπόν με τον τρόπο που ξεκίνησα. Δηλαδή είμαι βαθιά πεπισμένη ότι καμιά φορά δεν χρειάζεται νέα νομοθεσία. Ίσως μπορούμε να συμπληρώσουμε τα κενά με καλύτερη συνεργασία, δηλαδή με το να εμπιστευόμαστε τα εθνικά κοινοβούλια γιατί γνωριζόμαστε καλύτερα, γιατί εμπιστευόμαστε ότι κάνουν σωστά τη δουλειά τους σε τοπικό επίπεδο και να βελτιώσουμε και τη δικιά μας δραστηριότητα μέσω των οργανισμών που έχουμε καταρτήσει και στους οποίους έχουμε αναθέσει κάποια εντολή. ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα πριν αρχίσει η συζήτηση θα ακούσουμε την ακαδημαϊκή σκοπιά του, κυρίου, του καθηγητή Ορί Λαμπάη του Πανεπιστημίου της Μπαγιών. Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την πρόσκλησή σας και για την τιμή που μου κάνετε στην ανταλλαγή αυτή απόψεων με τους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Έχει περάσει η ώρα και γι' αυτό θα τα πω απλά χωρίς να υπησέλθω στις νομικιστικές λεπτομέρειες που χρησιμοποιούν διπλή γλώσσα για να αποφύγουν τις δυσκολίες. Θα μιλήσω λοιπόν ειλικρινά και όχι ακαδημαϊκά. Πρώτον, γιατί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση με την οποία δημιουργείται ο Ευρωπαϊκός Νομικός Χώρος. Σχεδόν 10 χρόνια μιλάμε για τη δημιουργία της ενίας αυτής, το 2002, 8 χρόνια. Και έχουν γίνει, έχει υποθεί ό,τι μπορούσε να υποθεί Ήδη από το 2003-2004 ως αντιρρήσεις ή διευθετήσεις τίποτα δεν έγινε εκ τότε. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε. Ποια μπορεί να είναι η διευθετησεις τιποτα δεν εγινε εκ τι μπορουμε λοιπον να κανουμε ποια μπορει να ειναι η αποτελεσματικοτητα που να αναμένουμε. Το 2002 ελήφθη μία το, απόφαση το Δεκέμβριο του 2008 μια δεύτερη και τίποτε άλλο. Το πρόγραμμα της Στοκόλμης ήταν μια στρατηγική για την εσωτερική ασφάλεια της οποίας η ανεπάρκεια για ήταν προφανής παρόλο το ότι η Κομισιόν ε, έλεγε ότι θα το εφαρμόσει. Διαπιστώνω λοιπόν κάτι πολύ απλό. Δεν αρκεί να γράφουμε όπως λέει η Κομισιόν ότι πρέπει να ενδυναμωθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στη δικαστική Ευρώπη. Πρέπει να εφαρμοστεί κιόλα. Πρέπει να φανεί ότι είναι και ωφέλιμη για την καθημερινή ζωή των πολιτών και της Ένωσης και πρέπει να βασιστούμε απλώς και μόνο στην ισχύουσα συνθήκη. Αυτό ξέρει να κάνει ένας καθηγητής δικαίου. Να συγκρίνει με την ομολογία και γι' αυτό εγώ ως νομομαθής χάνομαι όταν ακούω έννοιες όπως πολιτικό κύκλο, στρατηγικό πρόγραμμα. Τι είναι στρατηγικό πρόγραμμα, αυτά είναι έννοιες που ακούγονται από τις εταιρείες αξιολόγησης της Αμερικής. Αλλά το πρόβλημα, το ίδιο το πρόβλημα της καταπολέμησης της εγκληματικότητας είναι πανάρχαιο. Η προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων αλλά και των ενόχων επίσης. Επομένως τρεις απλές ιδέες. Πρώτον, να στηριχθούμε στη συνθήκη που μας τα λέει όλα. Τη συνθήκη της Λασαβόνας εννοώ. Γιατί σήμερα αυτό που ισχύει ακόμη του Άμστερνταμ. Δεύτερον, να δούμε αυτά που είπατε και εσείς κυρία μου προηγουμένως ότι οι κανονισμοί δηλαδή μπορούν να ενεργοποιήσουν την Ευρωτζούστ και τρίτον να δούμε ποια θα μπορούσε να είναι η διοκτική αρχιτεκτονική της Ένωσης πρώτον η λισαβονοποίηση της Ευρωδίκ, της Ευρωτζάστ δεν χρειάζεται γιατί η νομοθεσία βασίζεται στην απόφαση πλαίσιο του 2002 όπως τροποποιήθηκε το 2008. Αλλά αυτά σαν να μην υπήρχε η συνθήκη της Λισαβόνας. Δηλαδή με υπερβολική φρόνηση. Δεν μπορούμε πάντως να πούμε ότι έγινε καμία φοβερή επανάσταση με τη Λισαβόνα ως προς τα θέματα της δίωξης και της επιβολής του νόμου. Το κεφάλαιο 4 της συνθήκης θεωρεί ότι είναι θέμα συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ κρατών και δεν είναι θέμα ενωσιακό και αποκλειστικής διαδικασίας αλλά θέμα απλώς συνεργασίας μεταξύ κρατών που στηρίζει και καθοδηγεί η Ένωση. Παρά την κατάργηση των διακυβερνητικών πυλώνων. Άρα καταλήγουμε στο απλό συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκή διοίκηση δικαστών, δικαστική διοίκηση, ούτε δικαστική ολοκλήρωση. Οι εθνικές αρχές είναι πάντα οι αρμόδιες και πριν και κατά τη διάρκεια και μετά. Είναι απλή δομική συνεργασία όπως είπε και ο κύριος Βίλιαμς με στόχο να υπάρξει μια απλή διαμεσολάβηση μεταξύ ευρωπαϊκού και εθνικού επίπεδου, η οποία όμως είναι πολύ πολύπλοκη. Αν θέλουμε να καταλάβουμε το πρόβλημα πρέπει να πούμε αυτό, ότι όλα βασίζονται στην εθνική εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων. Και εδώ που είναι θέμα κυριαρχίας, δηλαδή το δικαίωμα της επιβολής κυρώσεων, η Ένωση δημιουργεί μηχανισμούς που αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιο δεσμευτικοί και αυστηρή από ό,τι αυτά που εφαρμόζουν τώρα τα κράτη-μέλη. Εξού και ότι εκφράζω τη λύπη μου γιατί η Ευρωτζούστ δεν εφαρμόζει, δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε, όσο θα έπρεπε, παρά την πρωτοτυπία των δομών της. Δηλαδή, αν πάρουμε τη συνθήκη, ο πιο ευνοημένος αυτός που τους κέρδισε όλους, δεν αναφέρω τους ειτημένους, είναι η Eurojust. Ο μοναδικός θεσμός δηλαδή που φαίνεται σαν ο κύριος μοχλός της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας είναι η Eurojust. Εξού και η το ενδιαφέρον για το άρθρο 85 της συνθήκης που θα έπρεπε αύριο, θα μπορούσε αύριο να μας επιτρέψει με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και καλύτερο συντονισμό καθώς και με στήριξη πάνω στους εθνικές δομές να δημιουργήσει μεγαλύτερη συνεργασία γιατί σήμερα ο ρόλος που παίζει είναι απλώς ε, δεν είναι δεσμευτικός είναι συμβουλευτικός αύριο βέβαια μας λέει η πρώτη παράγραφος ότι πρέπει να στηρίξουμε την Eurojust, αλλά η δεύτερη παράγραφος λέει να ενισχυθεί η συνεργασία και ο συντονισμός απλώς. Άρα, δεν καταλαβαίνουμε γιατί υπάρχει αυτή, αυτός ο δισταγμός για το άρθρο του 14. Καταλαβαίνουμε γιατί το κάνει το Συμβούλιο, αλλά δεν καταλαβαίνουμε γιατί τηρεί τέτοια στάση η Κομισιόν. Και εδώ είναι η δεύτερη ιδέα που θέλω να σας εκφράσω έχετε μία ιστορική ευθύνη τεράστια. Διότι όταν το άρθρο 95 αρχίσει να εφαρμόζεται δια της συνήθους νομοθετικής μεθόδου, όπως λέει δεύτερο, δεύτερο δάφιό του, θα χρειαστεί να ορίσετε και να καθορίσετε ορισμένα πολύ βασικά για το μέλλον του δικαστικού χώρου στην Ευρώπη. Δηλαδή τη δομή του, τη λειτουργία του, το, εύρος, το πεδίο εφαρμογής του και τα καθήκοντά του. Αυτά. Όλα αυτά. Και με βάση τρεις ιδέες. Ποινική δίωξη από εθνικές αρχές, συντονισμός των ερευνών, ενίσχυση της δικαστικής συνεργασίας, καθώς και ενισχυμένη με συνεργασία επίλυση διαφορών. Επομένως, ο Ευρωπαίος νομοθέτης πρέπει να σκεφτεί τρία πράγματα. Πρώτον, κάτι δομικό για να το πω έτσι, που μας οδηγεί να σκεφτούμε ποια είναι η δικαστοποίηση της Eurojust, που δεν είναι θεσμός σαν τους άλλους, γιατί αποτελείται κυρίως, όχι αποκλειστικά δυστυχώς, από από εισαγγελείς και δικαστάς. Θα παίρνει αποφάσεις που αφορούν τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Σε δομικό λοιπόν επίπεδο θα χρειαστεί να καθοριστούν ορισμένες προσαρμογές. Δηλαδή για να τα πω ομά, εγώ δεν είμαι πεπισμένος ότι είναι καλό πράγμα η μισθή των μελών του Eurojust να δίνονται από τα κράτη-μέλη από όπου προέρχονται. Δεν είναι αυτό καλή εγγύηση για την ανεξαρτησία τους. Ούτε εγγυάται το κριτικό τους πνεύμα. Έπειτα, τα δομικά προβλήματα. Ήταν τα δομικά προβλήματα αυτό. Δεύτερον, η Eurojust δεν έχει καταστατικό. Δεν μπορεί να μείνει ως έχει. Εδώ το θέμα δεν είναι η Ευρωδίκ να έχει δικαίωμα άμεσης έρευνας κλπ. καθόλου. Αλλά απλώς πρέπει να καταλάβουμε λειτουργικά ότι αν οι διώξει είναι θέμα των χωρών μελών παρόλα αυτά πρέπει να εφαρμόσουν τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει ελεύθερα γιατί έχουν εγκρίνει τη συνθήκη. Ακόμη και αν καθυστερούν, ακόμη και διστακτικά. Διαβάστε τη δήλωση 27 της διάσκεψης που έγινε για την συνθήκη της Λισαβόνας όπου τα εθνικά κοινοβούλια εκφράζουν τους δισταγμούς τους. Τεράστιους δισταγμούς. Τρίτη ευθύνη σας, πολύ καθοριστική, το αναφέρατε και εσείς κυρία μου, δεν θα πω πολλά, το θέμα της αξιολόγησης, διότι το τελευταίο εδάφιο του 95 το γράφει. Εδώ καθορίζουμε και τους τρόπους με τους οποίους θα συνδέονται το Ευρωπαϊκό και τα Εθνικά Κοινοβούλια με τις δραστηριότητες της Ευρωδίκ. Αυτό θέτει ορισμένα σημαντικά ερωτήματα. Όπως σας είπα η Ευρωδίκ δεν είναι όργανο σαν τα άλλα. Σας παρακαλώ. Στις 6.30 πρέπει να τελειώσουμε και έχουμε ακόμα και τις ερωτήσεις και τα λοιπά. Ναι, ναι. ναι όχι τρία λεπτά μόνο. Αποτελείται από δικαστάς και λόγω του διαχωρισμού των εξουσιών πώς θα ελέγχονται από τον νομοθέτη. Τέλος. Τέλος, η στρατηγική εσωτερικής ασφαλείας της Ένωσης, για την οποία γίνεται τόσος λόγος, αναφέρει τρεις φορές την Ευρωδίκ, άρα της δίνει μεγάλη σημασία. Και επαναλαμβάνω τώρα το επιχείρημα του Γιώργου Μόναρ που είχε πει «Από καιρού εις καιρών πρέπει να δεχόμαστε τις ήττες μας και η τελευταία έκθεση πεπραγμένων της Ευρωδίκ λέει ποιες είναι οι δυσκολίες. 1424 υποθέσεις. Ωραία. Αλλά είμαστε βέβαιοι ότι ο αριθμός αυτός είναι αντιπροσωπευτικός μιας βελτίωσης. Εγώ δεν είμαι καθόλου βέβαιος. Έπειτα. Ένα κράτος, ας μην πω πιο, ένα μεσογειακό νησί, δεν υπέβαλε ούτε μία υπόθεση στην Ευρωδίκ. Άρα πρόκειται για παράδεισο. Τρίτον, το Λουξεμβούργο και μόνο έθεσε περισσότερες επερωτήσεις από ότι ολόκληρη η Ισπανία. Δεν ήξερα ότι το Λουξεμβούργο ήταν Σικάγο. και η Ολλανδία τόσες υποθέσεις όσο και η Γαλλία. Εδώ η μία από τις δύο χώρες ή υπερβάλλει ή δεν υποβάλλει αρκετές υποθέσεις. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει ένας χώρος, ένα βήμα όπου να λέγεται ρητά ότι η αξιοπιστία της Ένωσης και αυτός ο χώρος ελευθερίας κλπ δεν είναι τόσο πρόβλημα αρχών όσο πρόβλημα αποτελεσματικότητας και προς τιμήν σας είναι που μας δίνετε αυτόν τον χώρο συζήτησης τουλάχιστον του προβλήματος. Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά για την ανάλυση σας και που επιταχύνατε στο τέλος την παρουσίασή σας. Αλλά είμαστε έτοιμοι τώρα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Έχω κάποια μέλη των κοινοβουλίων που θέλουν το λόγο. Θα ακούσουμε πρώτα τα μέλη των κοινοβουλίων και κατόπιν θα ξαναδώσουμε το λόγο στα μέλη του πάνελ για να απαντήσουν. Η κυρία Ταλενφίνα από το Συνδικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. είμαι συνάδελφοι, καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο και την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για αυτό το πολύ ενδιαφέρον απόγευμα που περάσαμε. Θεωρώ πολύ σημαντικό εμείς ε, να συναντιόμαστε μεταξύ μας ως βουλευτές είτε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είτε των Εθνικών Κοινοβουλίων να έχουμε τη ε, δυνατότητα να συζητούμε σημαντικά θέματα. Νομίζω ότι αυτό είναι ζωτική σημασία ε, τώρα. Η καταπολέμηση του διεθνού εγκλήματο απαιτεί και διεθνή συνεργασία οι εθνικές αστυνομικέ και δικαστικέ αρχές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται σε μεγάλες έρευνες που αφορούν πολλές χώρες. Στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι πρέπει να υπάρχει εξισορρόπηση μεταξύ των μέτρων της πρόληψης του κλίματος και μέτρων προστασίας των δικαιωμάτων του ατόμου η Eurojust και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο έχουν αποκτήσει ένα, ένα και σημαντικότερο ρόλο στις προσπάθειες να βελτιωθεί η συνεργασία στον τομέα του ποινικού δικαίου. Και ορισμένα από τα παραδείγματα που παρουσίασε ο κύριος Williams είναι πολύ σημαντικά. Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε τι προσπάθειε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη βελτίωση τη συνεργασία ε, στον τομέα του ποινικού δικαίου. Ταυτόχρονα πρέπει να διευκρινίσουμε ποιε θα έπρεπε να είναι οι αρχέ των εθνικών αρχών και τι μπορεί να εφαρμοστεί πιο αποτελεσματικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εδώ θέλουμε να τονίσουμε τον κεντρικό ρόλο της διακυβερνητικής συνεργασίας με τη Eurojust. Κατά την άποψή μας, αυτό το επίπεδο συνεργασίας ε, θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω. Ένα γραφείο, Ευρωπαϊκό Εγγελικό Γραφείο, δεν θα, ε, έχει, δεν θα είναι σε καλύτερη θέση να λύσει περαιτέρω προβλήματα συνεργασίας. Επίσης, είναι σημαντικό να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα των μέτρων που έχουν αποφασιστεί στο παρελθόν, προκειμένου να καθορίσουμε αν ε, εξυπηρετούν το στόχο τους θα πρέπει να ακολουθήσουμε την οδό που έχει θετηθεί και να ενδυναμώσουμε την αμοιβή εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών. Η βάση της συνεργασίας είναι η αρχή της αμοιβή αναγνώρισης των αποφάσεων σε ποινικά θέματα. Αυτό είναι ένα καθήκον το οποίο χρειάζεται χρόνο για να υλοποιηθεί. Και στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη τα μεμονωμένα νομικά συστήματα των κρατών μελών ε, και το σεβασμό των θεμελιωδών εθνικών αρχών του ποινικού δικαίου. Για το λόγο αυτό θα ήθελα και πάλι να τονίσω τη σημασία της διακυβερνητικής συνεργασίας με το Eurojust ιστορικό της Eurojust και αύριο στην ε, καταληκτική συνεδρίαση θα επανέλθω στο θέμα του κοινοβουλευτικού ελέγχου και της Europol και της Eurojust. Ευχαριστώ πολύ. Βλέπω να ζητούν και άλλοι το λόγο. Θέλω λοιπόν να σας υπενθυμίσω ότι πρέπει να σεβαστούμε τα χρονικά όρια. Πρέπει να ολοκληρώσουμε μέχρι τις 6.30. Ε, η κυρία Βασιλική Τσονόγλου από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ βεβαίως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι μεγάλη μου τιμή να τοποθετούμε, ε, ειδικά σε μια κρίσιμη για την πατρίδα μου περίοδο ε, είναι γεγονός ότι η διαφθορά έχει διωγγωθεί και ε, πράγματι τα επιχειρηματικά συμφέροντα που, μπαίνουν, που τείνουν να υπερκεράσουν την πολιτική πολλαπλασιάζονται. Συν αυτών βεβαίως είναι και η εγκληματικότητα η οποία αυξάνεται εν ώψη της κρίσης σε επίπεδα τα οποία ε, πράγματι έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα αλλά και σε αυτά τα οποία συμμετέχουν και άτομα που δεν υπάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Eurojust είναι πραγματικά ε, μια δομή η οποία ε, βοηθά τα εθνικά κοινοβούλια, τις εθνικές νομοθεσίες, τις εθνικές ποινικέ τουλάχιστον διώξεις. Θέλω να ρωτήσω αν είναι πράγματι στους στόχους και στις προτεραιότητες ώστε να υπάρχουν ειδικά ειδικά εκπονημένες ε, μελέτες ή αν υπάρχει ένας μόνιμος μηχανισμός ο οποίος θα εξετάσει πού συμπίπτουν οι νομοθεσίες των ε, κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν υπάρχει πρόθεση κωδικοποίησης των ποινικών ε, νομοθετημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την μορφή που ε, έχουν ενσωματωθεί στα εθνικά ε, συντάγματα δίκαια και αν πράγματι μέσα στους στόχους της Eurojust είναι και ο έλεγχος της εκτέλεσης των αποφάσεων που εκδίδονται μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά δηλαδή εκτέλεση αποφάσεων παραδείγματος χάρη επί επιμέλειας ανηλίκων και ούτω καθεξής και τέταρτον, πώς επιλαμβάνεται η Eurojust όταν υπάρχει ε, δίωξη συμμετόχων ε, ατόμων που δεν υπάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μελών, δηλαδή ε, κρατών μελών που δεν υπάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λυπάμαι, έθεσα πολλά ερωτήματα. Συμφωνώ με την τοποθέτηση ιδίω του τελευταίου ομιλητή του αξιότιμου κυρίου Λαμπάη και θέλω να δω πράγματι αν υπάρχει και ουσιαστική στις προθέσεις και στις προτεραιότητες αν υπάρχει και δικαιοδοτική πρόθεση δικαιοδοτικής ε, ε, ε, ε επίτευξης και του χαρακτήρα αν πράγματι δηλαδή θα φτάσει σε σημείο ποτέ η Eurojust να αποδίδει και δίκαιον. Ευχαριστώ. Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η κυρία Κίνγκα Κόνς. Ευχαριστώ. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο και ερώτημα. Ε, αναφερθήκαμε ε, το, ε, στην ε, Ευρωπαϊκό Ένταλμα Προστασίας. Πιστεύετε ότι βάσει αυτού του εντάλματος θα μπορέσουν οι εθνικές αρχές να συνεργαστούν πιο στενά και πιο αποτελεσματικά και να υπάρξει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη αμοιβαία από ό,τι στο παρελθόν. Επίσης η Eurojust μπορεί να επεξεργάζεται ορισμένα προσωπικά στοιχεία. Άρα δημιουργούνται ορισμένα ερωτηματικά σχετικά με την δημοκρατική ε, εξέταση ε, και σχετικά με το naming and shaming θα χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο στο μέλλον και τώρα από, το Ιταλικό, από την Ιταλική Γερουσία ο κύριος Αλμπέρτο Μαϊντάι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Τηλεγραφική παρέμβασή μου. Όμως πρέπει να κάνω δύο πολύ σύντομα σχόλια. Τώρα, σας υπόθηκαν από τη συνάδελφο από την Ελλάδα, δηλαδή, τι γίνεται με τη συνεισφορά μας ε, Δηλαδή πρέπει να ξέρουμε αν ανοίγει ένας διάλογος ε, μεταξύ μας ε, διαφορετικά η παρουσία μας εδώ σε καιρούς κρίσης γιατί αυτό κοστίζει ε, σε κάθε φορολογούμενο πολίτη αρχίζει να είναι προβληματική. Έτσι λοιπόν εμένα θα μου άρεσε να ξέρω αν αυτά που, εμάς, που εμείς προτείνουμε δεν λέω τέλος πάντων να γίνονται αποδεκτά αλλά αν λαμβάνονται υπόψη και με ποιους όρους. Λοιπόν, το δεύτερο σχολείο έχει να κάνει με όσα υπόθηκαν από την κυρία Αλφάνο, δηλαδή την αναγκαιότητα κατά την άποψή μου το Ευρωπαϊκό ε, Συμβούλιο να αποκτήσει, αν ε, όχι μία μόνιμη, μία προσωρινή εφήμερη επιτροπή όπου θα συμμετέχουν αρμόδιοι ε, περιγνώμονες που μπορούν να αξιολογούν τα τις διασυνοριακές εγκληματικές ε, ομάδες, τα φαινόμενα αυτά. Εμείς ε, ξεκινάμε από αυτό το δεδομένο. Έχουμε ένα φαινόμενο σε επέκταση στην Ευρώπη. Το πρόβλημα της μαφίας δεν είναι πλέον εθνικό, αλλά διεθνές. Τι κάνει η Ευρώπη συγκεκριμένα για να αποθήσει αυτή την επίθεση κατά των λευθυρών των πολιτών και Πρέπει να είμαι πολύ συνοπτικός. Ε, μιλάμε και για την Ευρωπόλ και για την Eurojust. Ε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για το ένα χωρίς να μιλήσουμε για το άλλο, γιατί ε, υπάρχουν ουσιαστικά μιλάμε για τις δύο ψήσεις του ίδιου νομίσματος. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για την Eurojust χωρίς την Europol. Έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ, Πρόεδρε, γιατί εδώ και χρόνια εμείς περιστρεφόμαστε γύρω από τι μπορούν να κάνουν οι Europol και οι Eurojust. Πριν λίγο ακούσαμε κάποιον που είπε τι ε, αν μπορεί να υπάρξει και νομολογία, αλλά με ποιο τρόπο εμείς πρώτα απ' όλα πρέπει να καθορίσουμε τα καθήκοντα της Eurojust. Δηλαδή είναι πολύ σοβαρό να μιλάμε εδώ για τη Eurojust και να λέμε ευρωδίκ χωρίς να έχει δικαστές. Είναι σοβαρή αντίφαση αυτό και μα είπατε έχετε 45 εισαγγελίε. Δεν καταλαβαίνω όμω ποια είναι η αρμοδιότητα των ανθρώπων αυτών και των υπόλοιπων 200 και των εμπειρογνωμόνων. Έχουμε λοιπόν ένα οργανισμό ε, και ο εκπρόσωπο ε, του οργανισμού αυτό είπε είναι μικρό αλλά πάρα πολύ αποτελεσματικό. Εγώ έχω κάποια αμφιβολία για την αποτελεσματικότητα. Όχι βέβαια ε, για αυτού που τον δικούν αλλά για τη δομή του οργανισμού. Λοιπόν, Ελπίζω να σεβαστώ και το χρόνο. πρέπει να κάνουμε και κάποιε προτάσει, γιατί δεν θα διαφορετικά να παρεμβαίνουμε. Πρέπει να παρέμβουμε έτσι ώστε να δώσουμε συγκεκριμένα καθήκοντα στην Γεροπόλ και στη Ζουρτζά. Δεν μπορούν να έχουν απλώ το σκοπό του συντονισμού αυτοί οι δύο οργανισμοί. Πρέπει να είναι χρήσιμοι αυτοί οι οργανισμοί. Πρόσωπο τη Eurojust μα είπε, ελπίσουμε, ότι θα στρέφονται σε εμά, θα απευθύνονται σε εμά όλο και περισσότερο τα κρατη Δεν μπορούμε. Ε, να πράξουμε κάτι τέτοιο μόνο μια πρόβλεψη. Ε, πρέπει να είναι χρήσιμο ο οργανισμό αυτό. Πρέπει να έχει μια βάση δεδομένων, πρέπει να έχει ουσιαστικά καθήκοντα και ουσιαστικέ γνώσει και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να στέλνουν τα στοιχεία του σε αυτή την βάση δεδομένων ε, όπως ε, έγινε και ε, κατά το Ιταλικό παράδειγμα έχουμε βάσεις δεδομένων για τη μαφία παραδείγματο χάρη και τοπικές που στέλνουν τα στοιχεία και συνδέονται με την κεντρική βάση δεδομένων. Εγώ ήθελα να καταθέσω εδώ αυτή την ανησυχία μου πρόεδρε. Δεν θα ήθελα η παρουσία μας εδώ ε, απλώς να παραμείνει κάτι τυπικό γιατί αν δεν μπορούμε να πούμε αυτό που εμείς θέλουμε να πούμε για να συνεισφέρουμε στον έλεγχο και στην ανάπτυξη. Αναρωτιέμαι γιατί ερχόμαστε τελικά εδώ. Ευχαριστώ. Από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, ο κ. Κωνσταντινός Σαβέρας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα εν πρώτης να συγχαρώ τον κύριο καθηγητή για το υψηλό επίπεδο των στοχασμών του και της κριτικής την οποία διατύπωσε, καθώς επίσης και να παραδεχτώ και εγώ και να ομολογήσω ότι πράγματι χρειάζεται ένα είδος γλωσσικής κάθαρσης σε πολλά κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να μπορεί ο καθένας από εμάς να αντιλαμβάνεται σε τι ακριβώς αντιστοιχεί στην πραγματικότητα ο κάθε όρος που χρησιμοποιείται γιατί πολλοί από αυτούς πάσχουν από μια αθεράπευτη μεγαλοστομία και κυρίως αναφέρομαι στην ίδρυση και τη λειτουργία του ενιαίου δικαστικού χώρου. Τι σημαίνει ενιαίος δικαστικός χώρος όταν είναι δεδομένο ότι την κυρίαρχη δικαιοδοσία, την αρμοδιότητα σε θέματα που έχουν να κάνουν με την απονομή του δικαίου την έχουν τα εθνικά κράτη. Και βεβαίως δεν μπορεί η οποιαδήποτε δραστηριότητα επάνω στο θέμα του ενιαίου δικαστικού χώρου δεν μπορεί παρά να περιορίζεται σε θέματα που έχουν να κάνουν με ζητήματα προδικασίας ή με ζητήματα εκτέλεσης αποφάσεων και ποινών. Αυτό όμως που έχει αξία να πούμε είναι ότι κάποια στιγμή ο πολίτης της Ευρώπης για να γίνει πραγματικά το επίκεντρο του ενδιαφέροντος αυτής της ευρωπαϊκής δημιουργίας θα πρέπει να αισθάνεται στην καθημερινή ζωή του τα αποτελέσματα της δράσης και της Europol και της Eurojust. Δυστυχώς όμως υπάρχει μια σειρά εγκλημάτων, τα ανάφερε προηγουμένως ο κύριος καθηγητής. Θα ήθελα μόνο να προσθέσω τα εγκλήματα διαφθοράς των πολιτικών και των κρατικών αξιωματούχων, στα οποία και η Europol και η Eurojust, όταν μάλιστα συμβαίνει να έχουν και διασυνοριακό χαρακτήρα που εμπλέκονται μεγάλα κράτη, μεγάλες ευρωπαϊκές δημοκρατίες, σιωπά, καθυστερεί ή, εν πάση περιπτώσει, δεν ανταποκρίνεται κατά τον τρόπο που οφείλει να ανταποκρίνεται. Επομένως, λοιπόν, καταλήγω, για να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε έλεγχο στη Eurojust ή να αξιολογήσουμε το έργο της, καθώς επίσης να την δεχτούμε σαν αποκλειστικά ωφέλιμο οργανισμό εργαλείο για τη δημιουργία του ενιαίου χώρου ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας θα πρέπει τουλάχιστον να πιστούμε ότι και από την σύστασή της και από τη λειτουργία της αλλά κυρίως και από την αποτελεσματικότητά της παράγει ωφέλιμο έργο για τον κάθε Ευρωπαίο φορολογούμενο πολίτη. Ευχαριστώ και τώρα μία τελευταία ερώτηση αλλά θέλω να σας πω ότι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μία εξήγηση είναι είναι μόνιμη κατάσταση και βασικός παράγοντας στην εργασία μας ο χρόνος. Λοιπόν, το σύστημα διερμηνίας πρέπει να λήξει στις 6.30. Έχουμε ένα πολύγλωσσο κοινοβούλιο και πρέπει πάντοτε να σεβόμαστε το χρόνο. Εδώ βέβαια πρέπει να αξιολογήσουμε το Eurojust, το Europol. Θα μπορούσαμε όλοι ο καθένας από εμά να σχολιάσει επί ώρες το θέμα αυτό, αλλά πρέπει να περιοριστούμε σε λίγες ερωτήσεις για να μπορέσουν να ε, απαντήσουν ε, οι θα είμαι πολύ σύντομο, Πρόεδρε, λέει ο κύριο Κροτσέτα. Θέλω να υπογραμμίσω ένα-δυο ζητήματα που προέκυψαν άλλωστε και από τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων. Το θέμα του ρόλου της Eurojust. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με το λόγο που πρέπει να πτυξούμε εμεί εναντί τη Eurojust, αλλά εγώ νομίζω ότι εμεί πρέπει να εξετάσουμε και όλη την νομοθεσία εσωτερικών υποθέσεων και δικαιοσύνη, γιατί προφανώ υπάρχει μια παραμόρφωση επί θεμάτων και επί προσεγγίσεων. Και φυσικά κάτι τέτοιο εξαρτάται από τα διάφορα κράτη τη μεταχείριση την χάνει κάθε υπόθεση, ενώ ε, η εγκληματικότητα αναπτύσσει όλο και περισσότερες σημαντικές διασυνδέσεις μεταξύ της. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Ε, εγώ, συγγνώμη, το, το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Ερευνών διορθώνει ο θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ χρήσιμο γιατί μας επιτρέπει να προχωρήσουμε. Αυτό, αυτή η εντολή ε, η ερευνητική συνίσταται στο εξή. Ε, Παραδείγματο χάρη, σύμφωνα με ε, το σχέδιο του Συμβουλίου, σε μία εντολή μπορεί να φύγει από ένα αστυνομικό τμήμα κάποια χώρα, γιατί μια ερευνητική εντελή εκδίδονται, παραδείγματο χάρη, ε, από δικαστέ και να εκτελεστεί από μια άλλη αστυνομική αρχή σε μια άλλη χώρα. Και αυτό γίνεται πάντοτε με το σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών. Και του αντικειμένου τη έρευνα, του πολίτη που είναι αντικείμενο τη έρευνα. και ε, ίσως ε, μπορεί η Eurojust να αναλάβει μεγαλύτερο ρόλο για να αξιολογεί μια τέτοια ιδέα έρευνα. Αυτό πρέπει να το σκεφτούμε. Και τελευταίο σχόλιο. Εγώ πιστεύω ότι δεν ε, ε, είναι πρόβλημα μόνο της Eurojust ότι δεν μπορεί να ξεκινήσει κάποια έρευνα. Αλλά το πρόβλημα ότι κάποιες χώρες δίνουν στοιχεία και κάποιες άλλες όχι, εδώ πρέπει να το δούμε αυτό το θέμα και πρέπει να εργαστούμε και με συγκεκριμένε εκθέσει. Πρέπει να δώσουμε αρμοδιότητα πρωτοβουλία στο Eurojust. Γιατί αν προσδώσουμε αυτά τα δύο, δηλαδή την εντολή έρευνα και την δυνατότητα, την αρμοδιότητα ε, πρωτοβουλία στη Eurojust, ε, τότε μπορούμε, το χάρη, να ξεπεράσουμε πολλές καταστάσεις ε, όπου έχουμε αντιστάσεις σε διάφορες χώρες. Σας υπενθυμίζω ότι οι διερμηνείς μας έδωσαν μερικά λεπτά ακόμη, αλλά είναι έτοιμοι να φύγουν, οπότε να είστε πολύ σύντομοι. Ευχαριστώ. Θέλω να αναφερθώ σε δύο θέματα. Πρώτα για την προστασία δεδομένων. Δεν θα μπορέσω να απαντήσω σε μεμονωμένες ερωτήσεις, αλλά σχετικά με την προστασία δεδομένων δεν νομίζω ότι πρέπει να ανησυχείτε για δύο λόγους, διότι τελικά ο κάτοχος της, της πληροφόρησης είναι το κράτος μέλος είτε μεταβιβάστηκε στην Europol ή στην Eurojust. Το κράτος είναι κάτοχος και ελέγχει τις πληροφορίες αυτές και η, ε, η δίωξη θα γίνει σύμφωνα με τον Εθνικό Δικαστικό Έλεγχο ε, υπό τον εθνικό έλεγχο. Οπότε και η ουσία του Eurojust είναι ότι υπάρχει δικαστική εποπτεία στα θέματα της Eurojust. Επίσης άκουσα και τις κρίσεις οι οποίες ε, εκφράστηκαν κατά της Eurojust. Πρέπει να σας πω ότι δεν δέχομαι πολλά από αυτές τις κρίσεις διότι ε, πρέπει να σας πω ότι η Eurojust τα 10 χρόνια χρόνια που υπάρχει ήταν μια αρκετά επιτυχής οργάνωση διότι βοηθάμε ε, τους ε, εισαγγελείς, τους ερευνητές και ε, επανέρχονται προς εμάς και αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να μεταβιβάσουμε τις εμπειρίες που έχουμε διδαχτεί και να θεωρηθούμε σαν ένα κέντρο εμπειριών για το μέλλον. Ευχαριστώ. Η κυρία Βέμπερ. Μία πρόταση. Εάν όντως θέλουμε να έχουμε έναν χώρο ελευθερίας και ασφαλείας στην Ευρώπη θα πρέπει στο μέλλον το Eurojust να είναι αναβαθμισμένο σε σχέση με σήμερα. Καταρτίστηκε πριν 10 χρόνια και σιγά σιγά και με την ε, έλλειψη εμπιστοσύνης από τα κράτη-μέλη τώρα τελευταίως βελτιώθηκε διότι έχει επιτύχει μέχρι στιγμής. Αλλά βεβαίως το Συμβούλιο οι κυβερνήσεις είναι αυτές οι οποίες διστάζουν περισσότερο να αναβαθμίσουν τις εξουσίες της Eurojust και να προχωρήσουν στο επόμενο επίπεδο δραστηριότητας. Ευχαριστώ ο κύριο Σαλαμπέη. Ε, μία λέξη και έναν αριθμό. Μία λέξη όσον αφορά τις προτεραιότητες των κατασταλτικών αρχών και πρέπει να το πω σε εσά εθνικούς βουλευτές ε, ε, σύμφωνα με το άρθρο των συνθήκων από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δηλαδή τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Ένας ε, αριθμός στη σελίδα 60 της εκθέσεως του Eurojust για το 2010 βλέπετε σε ένα σκαρίφημα πώς απεικονίζουν την κατάσταση και θεωρώ ότι είναι μία εξαιρετική οργάνωση η καρδιά της μελλοντική δικαστικής Ευρώπης που χρειάζεται τη βοήθειά σας για να αναπτύξει τις δυνατότητες τις οποίες της επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Συνθήκη. Ευχαριστώ ε, και σας υπενθυμίζω ότι αύριο το πρωί ε, θα ε, προεδρεύσει ο επικεφαλής ενός εθνικού κοινοβουλίου Κοινοβουλίου ο Λόρ Χάνι αύριο το πρωί και από το Λόρ ε, Χάνι of Chiswick και ε, θα ήθελα να σας πω ότι πρέπει να ε, έρθετε λίγο πιο νωρίς για να μπείτε μέσα στο κτίριο οπότε αύριο ε, θα υπάρχει ένα άτομο στην είσοδο όπως και σήμερα το απόγευμα για να σας υποδεχθεί και να σας προωθήσει και τώρα υπάρχει ένα κόκτειλ στην, στο δεύτερο όροφο στο κτίριο ΡΙΣΠΑΚ και σας προσκαλώ ε, για να έρθετε σε αυτή τη δεξίωση. Σας ευχαριστώ και θα σας δω αύριο το πρωί.